Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Επειδή η αντιπρόεδρή μας σήμερα δεν είναι διαθέσιμη και υπήρξε πρόταση να προεδρεύσω εγώ, απλώς να ρωτήσω αν υπάρχουν αντιρρήσεις. Εάν όχι, μπορούμε να προχωρήσουμε να δούμε το σημείο 7, η πορεία των εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωμεσογειακής Συνέλευση. Πέρσι, η Επιτροπή μα ενέκρινε μια έκθεση ίδια πρωτοβουλία για τι εμπορικέ σχέσει με την Ευρωμεσογειακή περιοχή, η οποία καθορίζει πω η εμπορική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για την όλη περιοχή που εκδημοκρατίστηκε με την Αραβική Άνοιξη πρέπει να συνεχιστεί. Θα δούμε λοιπόν από σήμερα ποια είναι η στατική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την όλη περιοχή προκειμένου να έχουμε διαρκείς και εντατικέ σχέσει σε διμερέ επίπεδο με συνολικέ ε, σχέσει ελεύθερου εμπορίου, αλλά και σε τομεακό επίπεδο με πρόσθετα πρωτόκολλα για τι υπάρχουσε ε, συμφωνίε σύνδεση που βρίσκονται από διαπραγμάτευση και με σκοπό να ενδυναμώσουμε και να δημιουργήσουμε μια ενιαία ελεύθερη περιοχή εμπορικών σχέσεων σε όλη την ε, ζώνη της Μεσογείου. Θα δούμε επίση τι γίνεται με τι χώρε με τι οποίε δεν έχουμε υπογράψει εμπορικέ συμφωνίε, όπω τη Λιβύη και τη Συρία. Και το τι γίνεται με την τραγική κατάσταση στη δεύτερη χώρα, τη Συρία. Εάν δεν υπάρξουν ε, εξελίξει, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα σχέδια τη επιτροπή για το μέλλον. Επειδή δεν υπάρχουν εδώ εισηγητές, να δώσω απευθεία το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Σοφία Μουνιώση είναι εδώ για να μας μιλήσει. Thank you. Um, σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη ικανοποίηση να έρχομαι να σας ε, ενημερώσω εδώ. Νομίζω η τελευταία φορά που συζητήσαμε τις σχέσεις ε, με τη Λατευτή της Μεσογείου στην Επιτροπή ήταν ε, το προηγούμενο καλοκαίρι όταν η Επιτροπή συζητούσε την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που υθετήθηκε στις ε, αρχές του φετινού χρόνου. Από πέρσι έχουμε διεξάγει πολλές προσπάθειες σε πολλά μέτωπα, όχι μόνο επί της διμερούς ε, στρατηγικής, αλλά και σε κάποια περιφερειακά θέματα. Δεν έχουμε μία συμφωνία, αλλά και με αυτούς ε, ε, αλλά υπάρχουν και κάποιοι με τους οποίους ε, δεν υπάρχει δυνατότητα να υπογράψουμε συμφωνία ελευθεροπορίου γιατί δεν είναι μέλη του ΠΟΕ. Θα ξεκινήσω καταρχήν με το πώς ε, έχει η κατάσταση για την προετοιμασία αυτών των FTA, των Συμφωνίων Ελευθερών Συναλλαγών και κατόπιν θα σας αναφέρω στο που βρισκόμαστε για την Πανευρωπαϊκή Σύμβαση, για τους κανόνες ε, καταγωγής και θα σας πω και κάποια λόγια για τη Συρία, την Αλγερία και τη Λιβύη, για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, οι Κομισιόν έλαβε διαπραγματευτικές οδηγίες ε, πέρσι το Δεκέμβριο από το Συμβούλιο. Αναμέναμε η διαδικασία αυτή να ήταν ταχύτερη. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι στις διαπραγματευτικές οδηγίες το Συμβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να υλοποιήσει μια διερευνητική, μια προπαρασκευαστική διαδικασία με κάθε ένα από τους εταίρους που εμείς θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί ήδη κατά τη διάρκεια του 2012. Ξεκινήσαμε διαδικασία με την Ισία, Μαροκό και ε, η Ορδανία το Μάρτιο. Στο στάδιο εκείνο η Αίγυπτος, που επίσης είναι πιθανός υποψηφίο, ε, δεν έδειξε ενδιαφέρον να δεσμευτεί σε αυτή την προπαρασκευαστική διαδικασία και ήρθαμε σε επαφή με τις χώρες αυτές, είχαμε συνεδριάσεις, ιδίως με την Τινησία και το Μαρόκο, όπου συμμετείχαν όλα τα Υπουργεία που θα συμμετείχαν στη συνέχεια στις διαπραγματεύσεις. Η ιδέα αυτών των προσκευαστικών συναντήσεων ήταν να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό οι χώρες αυτές ε, ήταν προώθημες και ικανές όχι μόνο να διαπραγματευτούν αυτές τις ε, συμφωνίες αλλά να εφαρμόσουν και τις μελλοντικέ ε, συμφωνίες και στην περίπτωση των μεσογειακών εταίρων η συμφωνία αυτή δεν θα επικεντρωθεί στην πρόσβαση στην αγορά γιατί ήδη έχουμε απελευθέρωση των ε, βιομηχανικών αγαθών και σημαντική απελευθέρωση για τα γεωργικά προϊόντα επίσης έτσι λοιπόν αυτές οι συμφωνίες θα επικεντρωθούν περισσότερο σε οικονομικά θέματα, θέματα διακυβέρνησης και σε ρυθμιστική σύγκληση προς το κοινοτικό κεκτημένο. Αυτή είναι τομείς που είναι δύσκολη κατά την άποψή μας για οποιοδήποτε εταίρο, καθώς απαιτείται απαιτούνται εσωτερικές μεταρρυθμίσεις σε ορισμένες περιπτώσεις και επίσης απαιτείται αυτοί να λάβουν ένα σαφή προσανατολισμό προ το κοινοτικό κεκτημένο. Κατά την παρασκευαστική διαδικασία σημειώσαμε καλή πρόοδο με την Τινσία και το Μαρόκο. Με την Ιορδανία η προπαρασκευαστική διαδικασία κάποια στιγμή μπλοκαρίστηκε, συναντηθήκαμε το Μάρτιο, αλλά από τότε δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία, γιατί ήθελαν να καλύψουν ε, στην σημερινή FTA και το θέμα των κανόνων καταγωγής. Εμείς ε, όμως θέλαμε να το καλύψουμε αυτό σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Με την Αίγυπτο απλά είχαμε κάποιες επαφές, τίποτα μας δεν έγινε. Με το Μαρόκο ολοκληρώσαμε την προσκευαστική διαδικασία στη Οκτωβρίου. και Επίσης παρουσιάσαμε μια έκθεση στην Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής και αυτό ήταν απέτηση στις διαπραγματευτικές οδηγίες, δηλαδή να γίνει μια διαβούλευση με την Επιτροπή βάση της έκθεσης της Κομισιόν. Αυτή η διαβούλευση ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή και τώρα απλώς προσπαθούμε να βρούμε ημερομηνίε για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο σε πολιτικό επίπεδο. Προσπαθούμε λοιπόν ε, να ορίσουμε πιθανές ημερομηνίε για τον Επιτροπή και τον ε, Μαροκινό Υπουργό και πιθανότητα θα συναντηθούν του χρόνου τον Ιανουάριο. Με την Τινησία είχαμε δύο συναντήσεις σε συνθήση Ολομέλεια τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο. Έχει προχωρήσει αρκετά η διαδικασία, αλλά πρέπει να την ολοκληρώσουμε. Χρειαζόμαστε μία ακόμη Ολομέλεια για να γίνει μια τεχνική δουλειά ακόμη και να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε μια έκθεση που θα παρουσιάσουμε στην Επιτροπή Εμπειρικής Πολιτικής. Τα καλά νέα από την ισιακή πλευρά είναι ότι κατορθώσαμε να έχουμε πολιτική επιβεβαίωση ότι ενδιαφέρονται για την DCFTA στη συνάντηση του Νοεμβρίου, στη συνάντηση του Συμβουλίου Σύνδεσης που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν ε, στα πλαίσια της προετοιμασίας αυτών των συμφωνιών. Πολύ σύντομα με το Μαρόκο θα ξεκινήσουμε αυτήν την προοπτική και με την Ισία θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προσκευαστική διαδικασία το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους και κάποια στιγμή στο πρώτο εξάμηνο του έτους θα μπορέσει να ξεκινήσει η συμφωνία με την Ιορδανία. Θα καθυστερήσουμε περισσότερο και χρειάζονται περισσότερες προετοιμασίες ε, πριν να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Παράλληλα με τις συμφωνίες αυτές συνεχίσαμε κάποιες διμερείς ε, διαπραγματεύσεις. Δεν σημείωσαμε ιδιαίτερη πρόοδο εκτός από τις διαπραγματεύσεις για τις υπηρεσίες με το Μαρόκο, αλλά ακόμη και στις διαπραγματεύσεις αυτές δεν ε, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις αυτές ακόμη και το πιο πιθανό σενάριο είναι να συμπεριληφθούν στις διαπραγματεύσεις για την DCFTA, αλλά λαμβάνοντας υπόψη το που έχουμε φτάσει σήμερα. Έτσι λοιπόν δεν θα ξεκινήσουμε από το μηδέν, απλώς θα συνεχίσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Είμαστε ετοιμοί να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, με την Τινησία για την ΑΚΑ, δηλαδή για την συμφωνία ε, με την ε, πρόσβαση στα βιομηχανικά προϊόντα και ουσιαστικά πρέπει να γίνει μια διαδικασία ολοκλήρωσης της νομοθεσίας από την και πλευρά. Έτσι λοιπόν και σε οριζόντιο επίπεδο και σε τομεακό επίπεδο για τους δύο τομείς που έχουν επιλέξει πρέπει να το πράξουν αυτό, αλλά αυτό δεν έχει λάβει χώρα ακόμη. Ελπίζουμε ότι αυτή την εβδομάδα ο Επίτροπο Ταγιάννη θα μεταβεί στην Τινησία και πιθανότατα θα πει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το τεχνικό έργο πριν να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Τινησία. Για τις ε, διαπραγματεύσεις για το γεωργικό τομέα, τα γεωργικά προϊόντα δεν ε, μας είπε με σαφήνεια η Τινησία και η πλευρά ότι θέλει να ξαναρχίσει αυτές τις διαπραγματεύσεις ή δεν μπορούσαν να λάβουν κάποια απόφαση μάλλον. Έτσι λοιπόν προς το παρόν δεν έχουν ξεκινήσει αυτές οι διαπραγματεύσεις εκ νέου και πιθανόν θα συμπεριληφθούν στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Σε περιφερειακό επίπεδο συνεχίζουμε να προωθούμε την αναθεώρηση των κανόνων καταγωγής ε, στο πλαίσιο της σύμβασης της ε, η οποία υπεγράφει πέρσι τον Ιούνιο. Δεν έχει όμως ε, επικυρωθεί ακόμα από καμία χώρα της Νοτιού Μεσογείου. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί η αναθεώρηση των κανόνων τελικά θα αποφασιστεί από αυτούς που έχουν κυρώσει τη σύμβαση. Και επομένως ασκούμε επίση στις ε, μεσογειακές χώρες να υπογράψουν γρήγορα και να προηγούν σε κύρωση. Η Μαρόκο και η Ορδανία έχουν υπογράψει, είναι στη διαδικασία της κύρωσης αλλά δεν υπάρχουν άλλες χώρες που να έχουν υπογράψει προς το παρόν. Θα χρειαστεί λοιπόν κάποιος χρόνος μέχρι να έχουμε ένα σοβαρό αριθμό εταίρων από την Νότια που να έχουν κυρώσει τη σύμβαση. Η διαδικασία αναθεώρησης προχωρά πολύ αργά, πολύ πιο αργά από ό,τι αναμέναμε αρχικά επειδή υπάρχουν αποκλίνουσες θέσεις των διάφορων ομάδων χωρών που συμμετέχουν στον χείρημα αυτό. Βλέπει κανείς ε, ότι η Τουρκία ή οι μεσογειακοί δεν ενδιαφέρονται στο ίδιο επίπεδο. για ορισμένες περιοχές, για ορισμένους τομείς, όμως ε, τους επόμενους μήνες δεν περιμένουμε να υπάρχουν εξέλιξεις σε αυτό το θέμα και περιμένουμε ότι το πρώτο εξάμεινο του 2013 θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό στους περισσότερους τομείς όπου μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και να απομονώσουμε του δύο-τρει πολύ δύσκολου τομεί, συμπεριλαμβανομένου και των πλώστο-εφαντουργικών. Αυτό θα είναι ένα από του πιο δύσκολου τομεί για να καταλήξουμε σε συμφωνία στο πλαίσιο αυτή τη σύμβασης. Γιατί υπάρχουν ε, πολύ διαφορετικέ θέσει, αν δείτε τη θέση τη Ιορδανία ή τη Τουρκία, λόγου χάρη. Επιπρόσθετα, η Κομισιόν συνεχίζει να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μηχανισμό εμπορίου, διευκόλυνσης εμπορίου και επενδύσεων για να βελτιωθεί το εμπορίο και οι επενδύσεις στη Μεσόγειο. Ολοκληρώνουμε τη σύνδεση με ένα διεθνή οργανισμό που θα υιοθετήσει το project. Επομένως, μάλλον θα υπάρχει από του χρόνου. Αυτό είναι καλό νέο για μας, γιατί είναι κάτι που λείπει οι οικονομικοί φορείς δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που διατίθεται στο εργαλείο αυτό, σε αυτό το μηχανισμό. Και να πω και δύο λόγια για τις άλλες χώρες με τις οποίες ε, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τέτοιου είδους ε, συμφωνίες, γιατί δεν είναι μέλη του ΠΟΗ. Η Αλγερία παραμένει ένα σημαντικός εταίρος για μας ακόμη και αν δεν είναι άμεσο υποψήφιο για μια DCFTA, βέβαια πρέπει να μπει στον ΠΟΕ. Οι διμερείς διαπραγματεύσεις για τον ΠΟΕ δεν είναι εύκολες. Η Αλγερία έχει μια δύσκολη στάση για τις υπηρεσίες τα προηγούμενα τρία-τέσσερα χρόνια έχει βάλει περιορισμούς στις επενδύσεις που τώρα έχουν συμπεριληφθεί στην διαδικασία πρόσβαση στον ΠΟΕ. Αυτό σημαίνει ότι παναχωρούν σε αυτό το τομέα. Έτσι λοιπόν δεν θα είναι εύκολη η διαδικασία, αλλά για μας παραμένει άμεση προτεραιότητα. Γιατί πιστεύουμε ότι με, χωρίς πρόσβαση στον ΠΟΕ δεν μπορούμε να σκεφτούμε μία εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων μια συσφίξη των εμπορικών σχέσεων. Οι Αλγερινοί όμω μα είπαν ότι θέλουν να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία. Διαπραγματευόμαστε ένα σχέδιο δράση μαζί του και στο σχέδιο αυτό θα υπάρχουν μέτρα για ρυθμιστική σύγκληση σε πολλού τομεί. Και αυτό είναι καλό νέο για μα. Η Αλγερία θα πρέπει δηλαδή να συμπεριλάβει τμήματα του κεκτημένου υπό το σχέδιο δράσης για τη Λιβύη. της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, οι προτεραιότητές τους αυτή τη στιγμή δεν είναι να ξαναρχίσουν οποιασδήποτε εμπορικές διαπραγματεύσεις. Δεν ε, κάνουμε λοιπόν ε, κάποια δραστικά βήματα για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Ε, οι διαπραγματεύσεις όταν συνεχίζονταν ήδη φαινόταν από τότε ότι ήταν πολύ φιλόδοξη συμφωνία για τη Λιβύη. Μάλιστα αποκλειόταν ότι ε, θα έχουμε μια τέτοια, ένα τέτοιο χώρο βαθύτερο συναλλαγών. Έτσι λοιπόν, θα μπορούσαμε να συνάψουμε κάποιε συμφωνίε με τη Λιβύη, αλλά δεν έχει έρθει ακόμη το πληρώμα του χρόνου. Αναφέρατε και τη Συρία. Η συμφωνία σύνδεση ε, μονογραφήθηκε και ε, μάλιστα αναθεωρήθηκε και το 2009. Η κατάσταση έχει ω εξή. Δεν επιδιώκουμε την υπογραφή αυτής της συμφωνίας όταν εξελιχθεί η κατάσταση, η συμφωνία σύνδεσης μπορεί να τεθεί εκ νέου επιτάπητος. Όμως προς το παρόν, δυστυχώς με τη Συρία, μάλλον ακολουθούμε το σενάριο όσο το δυνατόν λιγότερα και μάλλον επιβάλλουμε περιοριστικά εμπορικά μέτρα παρά προς το να κινηθούμε, κινούμαστε προς το να έχουμε περιοριστικά εμπορικά μέτρα παρά να έχουμε διευκόλυνση του εμπορίου. Αυτό συμβαίνει με τους κύριους εταίρους, με τους οποίους συνεργαζόμαστε ενεργά στη Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να δώσω το λόγο στους βουλευτές, ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε όσον αφορά τις ε, προσπάθειες της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής να συνάψει συμβάσεις με τις χώρες της Μεσογείου, αυτές τις προσπάθειες τις βρίσκω σημαντικές, κυρίως έχοντας κατά νου ότι οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις για την ενίσχυση της δημοκρατίας πρέπει να στηριχθούν Κατόπιν τούτου είναι σημαντικό να συναυθούν λογικές συμβάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν τι ακριβώς συμβαίνει με τους ε, εμπλεκόμενους. Δηλαδή, διαπραγματευόμεθα με τέρους, αλλά αυτό στηρίζεται από την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η δική μου εντύπωση είναι η εξής, ότι σε αντίθεση με τις ε, περιόδους ε, πριν από τη δημοκρατία, αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή οικονομία και η βιομηχανία δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη Μεσόγειο. Παραδείγματο χάρη, αν δούμε τις ε, επενδυτικές δραστηριότητες στην Αίγυπτο, διαπιστώνουμε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμη να προβεί σε επενδύσεις στην Αίγυπτο. Αυτό λοιπόν η Κομισιόν το επιβεβαιώνει ή όχι. Και κατ' ουσίαν πώς μπορούμε να μεριμνήσουμε έτσι ώστε παράλληλα με τις ε, διαπραγματεύσεις ε, να υπάρχει και μία άλλου είδους ε, οικονομική στήριξη έτσι ώστε και οι επιτόπιοι εταίροι να δραστηριοποιηθούν για να δημιουργηθούν ε, θέσεις απασχόλησης κυρίως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Νομίζω ότι το σκηνικό των δημοτεύσεων όπω είπε και ο Πρόεδρο, είναι η Αραβική Άνοιξη και εξελίξει στην Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Καλό είναι λοιπόν να θυμίσουμε, και ίσω αναγκαίο να είναι κιόλα, ότι υπό το φω αυτών των γεγονότων χρειάστηκε νέα προσέγγιση στο κοινό έγγραφο τη 27η Νοεμβρίου ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις σχέσεις με την ε, περιοχή της Μεσογείου. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κατά πόσον ε, υπάρχει αυτή η νέα προσέγγιση ακόμα. Αναφέρονται οι ανάγκη για δεσμεύσεις ελεύθερων ε, εκλογών, για ελεύθερες συγκεντρώσεις και έκφραση απόψεων για την ασφάλεια και το κάτω δικαίου και τις δυνάμεις καταστολής για την δικαιοσύνη και την ελεύθερη άσκηση της δικαιοσύνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει λοιπόν ότι μπορεί να προχωρήσει αλλά δεν ανησυχεί πλέον για τα ζητήματα αυτά όπως αναφέρονται στο έγγραφο της 20ης Νοεμβρίου με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Είδαμε με τον πρόεδρο Μόρση να υπάρχουν προβλήματα με τον κεντρικό χαρακτήρα που θέλει να δώσει στην εξουσία και το κατά πόσον είναι αυτόνομη η δικαστική εξουσία. Στην Ιορδανία βλέπουμε να μην υπάρχει καμία ελευθερία συγκέντρωσης και ούτε ελευθερία διαπραγματεύσεων. Αυτά είναι μέρημνες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της νέας προσέγγισης που είχε προαναγγείλει. και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των συμφωνίων ελευθερμπορίου και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να λάβει υπόψη τη μελέτη αντικτύπου βιωσιμότητα τη Ευρωμεσογειακή Ζώνη από το 2007, η οποία αναφέρει μια σειρά από αρνητικέ επιπτώσει σε σχέση με την αύξηση τη ανεργία, την ε, τις περικοπές τους μισθούς, την έλλειψη κυβερνητικών εισοδημάτων και την περικοπή δαπανών για τις κοινωνικές υπηρεσίες στις χώρες της Βορειοαφρικής. Τι προτείνει διαφορετικό αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς σκοπεύει να αποφύγει τις ε, αρνητικές αυτές συνέπειες της υλοποίησης των Συμφωνιών Ελευθερίου Εμπορίου. Uh, Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω και εγώ ένα δικό μου ερώτημα. Κοιτάξτε, ε, το 2010 είχαμε ως ε, στόχο να ολοκληρωθεί αυτός ο χώρος Euromed. Τώρα εντωμεταξύ έχει προκύψει η Αραβική Άνοιξη και έχει χαθεί η προθεσμία. Αν κατάλαβα καλά αυτά που μας είπατε, καταλήγετε στο ότι εσείς ε, ελπίζετε ε, να υπάρξει πρόοδος ε, με κάποιες μεμονωμένες χώρες, αλλά μία συνολική πρόοδος για τη Μεσόγειο, αυτό δεν το βλέπετε ε, να προχωράει. Δηλαδή, κατ' ουσίαν τι συμβαίνει, έχει πεθάνει αυτό το σχέδιο, μήπως ε, πρέπει να προχωρήσουμε με μονομένες χώρες ή είναι καλύτερα να περιμένουμε έτσι ώστε να προχωρήσουμε ε, με το σύνολο των χωρών. Και αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια από τα μέλη, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ξεκινήσω με την ερώτηση για τις επενδύσεις. Τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που είχα πει για τις επενδύσεις μας δείχνουν το αντίθετο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος επενδυτής στην περιοχή και προπορεύεται κατά πολύ και δούμε τις στατιστικές για την Αίγυπτο, για το Μαρόκο, για την Ισία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναλογεί περίπου από τα 2 τρίτα στο 90% των επενδύσεων στις χώρες αυτές για πέρσι. Είναι σαφές λοιπόν ότι εξακολουθεί να υπάρχει βιομηχανία και να ενδιαφέρεται για τις χώρες αυτές. Μπορεί το ενδιαφέρον να διαφέρει αναλογώς με τους τομείς και με τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κράτη-μέλη που είναι πιο παρόντα στην περιοχή αυτή από, τις, ε, από τη άλλα. Αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την ευρωπαϊκή βιομηχανία να εξελίψουμε τα μετασμολογικά εμπόδια, να υπάρχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς το επενδυτικό κλίμα. Και αυτά είναι τα κύρια στοιχεία που επιδιώκονται ε, στη σφαιρική και σε βαθοζώνη ελευθερών συναλλαγών. Όπως είπα, δεν είναι ένα θέμα πρόσβαση στην αγορά τόσο, είναι περισσότερο θέμα ρυθμιστικής σύγκλησης. Είναι αλήθεια ότι στην Αίγυπτο υπήρξαν πολλά προβλήματα από πέρσι με επενδύσεις στη χώρα και σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα δικαστήρια για τις προηγούμενες ιδιωτικοποίησεις, αλλά και επειδή υπήρξε μια σειρά μέτρων που υιοθέτησε πρόσφατα η Αίγυπτος, που δεν διευκόλυναν τη ζωή των εταιριών μας και αυτό είναι ένα γεγονός, γιατί αυξήθηκαν και τα μέτρα αυτά. Αυξήθηκε ο ρυθμός τους παράλληλα. Συνεχίζουμε να συζητούμε με τις Αιγυπτιακές Αρχές για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα πρόσβαση στην αγορά. Συνεχίζουμε να έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο μαζί τους. Ακόμη λοιπόν και αν η προπαρασκευαστική διαδικασία για τι διαπραγματεύσει θα μπορούσε να καθυστερήσει, να χρειαστεί περισσότερο χρόνο στην περίπτωση του Αιγύπτου. Εμεί θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα και υπάρχει σήμερα και συμφωνία σύνδεση που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να συνεχίσουμε τι συζητήσει με την Αιγυπτιακή πλευρά για όλα τα μέτρα που εφαρμόζουν. Όμως γενικά εξακολουθούμε να βλέπουμε ενδιαφέρον από την ευρωπαϊκή βιομηχανία για τις χώρες αυτές. Στην περίπτωση του Μαρόκου είναι σαφές. Στην περίπτωση της Τινησίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος πρωταγωνιστής επίσης. Επομένως, βλέπουμε και μια ανάγκη να συνεχίσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις ως έναν τρόπο να προωθήσουμε και να διευκολύνουμε τις δραστηριότητες αυτών των επιχειρηματιών στις χώρες αυτές. Δεν έχουμε αλλάξει την προσέγγιση σε σχέση με τα όσα είπαμε πέρσι. Είναι σαφές ότι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, θα επιδιώξουμε κεφάλαια υφοροανάπτυξης και αυτό είναι τμήμα της συζήτηση που είχαμε με τις χώρες αυτές στην περοπαρασκευαστική διαδικασία. Για να σας αναφέρω το παράδειγμα του Μαρόκου, με το οποίο θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις. Μα έδωσε το Μαρόκο μια σαφή απάντηση. Θέλει να διαπραγματευτεί ένα κεφάλαιο για την αηφοροανάπτυξη και θα πρέπει να πιέσουμε το Μαρόκο για την ε, κύρωση της μόνης σύμβασης ΔΟΕ που δεν έχουν κυρώσει ακόμη μεταξύ των κυρίων συμβάσεων της ΔΟΕ. Είναι σαφές επίσης ότι σε όλες τις χώρες έχει αλλάξει η κατάσταση σε ό,τι αφορά στο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Αναφέρομαι τώρα πιο συγκεκριμένα στο Μαρόκο και στην Τινησία γιατί έχουμε προχωρήσει περισσότερο μαζί τους. Και στις δύο περιπτώσεις ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών έχει γίνει τώρα τμήμα των εθνικών πολιτικών και πρέπει στο διάλογο αυτό πρέπει να ελοποιείται ο διάλογος αυτός και για εγχώριες αλλά και για διεθνείς πρωτοβουλίες και αυτό το κεφαλοποιούμε σε όλες μας τις συμφωνίες. Όταν ε, λάβαμε τις διαπραγματευτικές οδηγίες πέρσι για τις CFTAs, η ιδέα ήταν, ε, όπως ισχύει ε, και για τους εταίρους εξανατολάς, να διεξαγάγουμε τις διαπραγματεύσεις και να εξετάσουμε τα δημοκρατικά κριτηρία τα οποία αναφέρατε τη στιγμή της σύναψης των συμφωνιών αλλά βεβαίως εξετάζουμε και το πώς εξελίσσεται η κατάσταση κατά τη διάρκεια της προπερισχρηστικής διαδικασίας. Και όπως είπατε, ε, μας ανησυχεί και εμάς, μας ανησυχούν και εμάς τα πρόσφατα γεγονότα στην Αίγυπτο και ε, τη εξέλιξη ακολουθεί κατάσταση. Όπως είπα, η διαδικασία με την Αίγυπτο θα καθυστερήσει. Αναφέρατε τις μελέτες αντικτύπου της βιωσιμότητας του εμπορίου. Ε, είχαμε μία μελέτη αντικτύπου που υλοποιήσαμε το 2007 και τοποθετήκαμε και το 2009 σχετικά. Θα υλοποιήσουμε νέες τέτοιες μελέτες αντικτύπου γιατί πιστεύουμε ότι έχει αλλάξει η κατάσταση κατά πολύ. Και οι συμφωνίε που θα διαπραγματευτούμε τώρα είναι πολύ συγκεκριμένε. Χρειάζεται λοιπόν μία νέα εκτίμηση. Κανονικά η διαδικασία θα ξεκινήσει πριν από τα τέλη του 2012. Θα υπογράψουμε μια σύμβαση το Δεκέμβριο λογικά και ελπίζουμε ότι τις μελέτες θα τις έχουμε διαθέσιμες του χρόνου το Σεπτέμβριο για το Μαρόκο και την Τινησία. Για την Αίγυπτο και την Ιορδανία θα είναι τον επόμενο χρόνο. Αλλά θα υπάρχει χρόνος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις. Πρέπει λοιπόν να δούμε πότε θα συναυτούν οι, συμφων... συμφωνίες και να λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα των μελετών αντικτύπου. Προς στιγμή να επικεντρωνόμαστε σε αυτές τις δημοτικές διαπραγματεύσεις, αλλά δεν ξεχνάμε την περιφερειακή διαδικασία. Δεν ανέφερα την υποστήριξη μας ε, στη Συμφωνία Κάδη το Γαντήρ είχαμε μια συνάντηση με τα μέλη φέτος το Σεπτέμβριο και συνεχίζουμε να Συζητάμε πώς θα βελτιωθούν οι περιφερειακές συμφωνίες, θα προσφέρουμε τεχνική βοήθεια τώρα στην Παλαιστινιακή Αρχή, που επίσης θα συμμετάσχει στη συμφωνία αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς. Η περιφερειακή ολοκλήρωση δεν γίνεται ε, πριν να υπάρξει διμερής ε, ολοκλήρωση. Έτσι λοιπόν ε, εμείς ε, θεωρούμε ότι καταρχήν διμερώς οι χώρες κάνουν πράγματα μαζί μας και κατόπιν ε, ουσιαστικά ακολουθούν την ίδια διαδικασία και στις πολυμερεί του σχέσει. Τουλάχιστον αυτό έχουμε δει μέχρι σήμερα. Και επίση οι σφαιρικέ και σε βάθο ζώνε ελευθερών συναλλαγών έχουν κάποια αποτελέσματα τα οποία διαδίδονται, γιατί από τη στιγμή που κάποιε χώρε έρχονται σε προσέγγιση με το κεκτημένο, με το κοινοτικό κεκτημένο, με του ίδιου κανόνε δηλαδή, ουσιαστικά εξελίφουν και τα εμπόδια και μεταξύ τους γιατί θα έχουν κάποια ρυθμιστικά πλαίσια σε ορισμένους τομείς που θα βασίζονται στις ίδιες αρχές. Επομένως, όλα αυτά προωθούν και την περιφερειακή ολοκλήρωση κατά την άποψή μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτή την επισκόψη. Γνωρίζετε ότι έχουμε δύο ομάδες, δύο monitoring ομάδες για, τα θέματα αυτά. Ο κ. Δεζάουνες είναι ο μόνιμος ε, εισηγητής για την ε, περιοχή αυτή. Και η γνωμοδότηση πρωτοβουλίας, πρωτοβουλίας ε, πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία πέρσι με εισηγητή τον κύριο Ρινάλντι. Thank you very much. If there are no other comments, then I would like to go to point Εάν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πάμε στο σημείο 8, αντιπροσωπείο στη Ρωσία. Προέδρευσε ο κύριος Μορέιρα από την Επιτροπή μας και επισκέφθηκε την Μόσχα στα τέλη Οκτωβρίου. Η αντιπροσωπεία εκπροσωπούσε τέσσερι πολιτικές ομάδες και βασικό σκοπός αυτής τη αποστολή ήταν να αποτιμήσει το μέλλον των εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωσης-Ρωσίας. Η Ρωσία μόλις έγινε μέλος του ΠΟΕ τον Αύγουστο μόλι φέτος και φαίνεται ότι θα υιοθετήσει νέε εμπορικέ προδιαγραφέ. Επίση, η διαπραγματεύση των νέων εμπορικών ρητρών τη Νέα Συμφωνία μεταξύ Ρωσία και Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε τελικά σε αδιέξοδο. Η αντιπροσωπεία είχε ειλικρινεί και ανοιχτέ σχέσει με την κρατική δούμα, την κυβέρνηση, εκπροσώπους ε, του επιχειρηματικού κόσμου, των ρωσικών συνδικαλιστικών οργανώσεων κ.ο.κ. Όμω ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί πρόοδο λόγω τη στάσης αδιαλαξία των Ρώσων. Υπάρχει το σχετικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τι εμπορικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία και θέλαμε να περάσουμε το μήνυμα ότι η, Ευρωπαϊκή, ότι η Ρωσία πρέπει να εκπληρώσει τι ε, επιχρεώσει τη σύμφωνα με τον ΠΟΕ και να άρει του εμπορικού φραγμού. Επίση, θέλαμε να υπάρξουν δεσμευτικέ διατάξει στη νέα συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία ιδίω στον τομέα τη ενέργεια ε, Κάναμε επίση προσπάθειε να δούμε τι γίνεται με τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την ενίσχυση τη Τελωνιακή Ένωση και το πώς ε, βλέπει η Ρωσία τη μελλοντική ε, ολοκλήρωση των σχέσεών της με τους δικούς της ε, γείτονες από εμπορικής σκοπιάς. Θα δούμε τώρα τις απόψεις των μελών που βρίσκονταν στην επίσκεψη αυτή. Υπάρχουν βουλευτές που θα ήθελαν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Λάγκ. Ο Λάγκε, μάλλον... Muchas gracias, señor presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα κατά πρώτον να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής αυτής για την διοργάνωση της επίσκεψης. Η επίσκεψη στη Ρωσία έχει ως βασικό σκοπό να γνωρίσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις της προσχώρησης της χώρας αυτής των ΠΟΕ μετά από 18 χρόνια διαπραγματεύσεων. Θέλαμε να δούμε ποιες είναι οι εμπορικές προτεραιότητες της Ρωσίας, ποιες είναι οι προοπτικές της στο πλαίσιο αναθεώρησης της, της ε, εταιρικής σχέσης εμπορικής συνεργασίας και βεβαίως και από δημιουργούς άποψης τι γίνεται. Συναντήσαμε εκπροσώπους όλων των ε, τομέων προτεραιότητας εκπροσώπους με κυβερνητικών οργανώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, οργανώσεων εργοδοτών, ενώσεων μάλλον εργοδοτών, κυβερνητικού εκπροσώπους της Ρωσίας. Θέλαμε να δούμε ποιε είναι οι περιοπικέ προτεραιότητε που απασχολούν αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω για παράδειγμα, ότι τα τελευταία χρόνια υιοθέτησε μέτρα η Ρωσία για τα ελαφρά οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, μας ανησυχούσαν οι αποφάσεις της για την δεσμολόγηση της ανακύκλωσης των εισαγόμενων οχημάτων μέτρο που αντίκειται ακριβώ στις αρχές του ΠΟΕ ή η απαγόρευση εισαγωγής ζώντων ζώων προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε ζητήματα που έθιξε ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά τη Ρωσία σε ό,τι αφορά το κόστος τέτοιων ε, μέτρων τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Στη Ρωσία δεν υπάρχει οργανωμένη μέση τάξη. Και σε ό,τι αφορά τις νέες, σχέσεις, τις νέες συμφωνίες εταιρικής σχέσης, αυτές δεν έχουν ε, το σωστό υπόβαθρο. Ο εκπρόσωπος του εμπορικού επιμελητηρίου έκανε κάποιε ενδιαφέρουσε παρατηρήσεις, ιδίω ό,τι αφορά την απαγόρευση εισαγωγής των ζώων και μπορέσαμε έτσι να έχουμε καταλλαγή απόψεων με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Μας είπαν ότι θα υποβληθούν προτάσει σε επίπεδο ΠΟΕ όμως και ότι ενδεχομένω να ληφθούν κάποιες αποφάσει πολύ σύντομα. Επίση υπήρξε συνάντηση με μέλη της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εταιριών που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. Υπήρξαν αποκλίνουσες απόψεις. Γιατί για κάποιου. Ε, κατά την άποψη κάποιων υπήρξαν εξέλιξεις, άλλοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πρόοδο στη Ρωσία. και ρώτησα ποια είναι η κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πώς επηρεάζονται στις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Μας είπαν ότι υπήρχαν τάσεις εξυγχρονισμού και αλλαγή της δομής των εταιριών αυτών. Η κατανάλωση της μέσης τάξης αυξάνεται. Υπάρχει ε, συνεχής αύξηση για τη διαφθορά μας είπανε ότι θίγει μόνο τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης μας ε, είπαν ότι υπάρχουν τρία προβλήματα για κανείς δεν θέλει να μιλήσει αυτή τη στιγμή γι' αυτό όπως είναι η εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή φεύγουν πάρα πολλοί νέοι για να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Ένα άλλο πρόβλημα που έβλεπαν ήταν το θέμα των υποδομών, το θέμα του νερού και της αποχέτευσης. Ε, είναι πάρα πολλά έξοδα αυτά για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις και επίσης το δημογραφικό πρόβλημα. Οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις μας είπαν ε, ότι πρέπει να τις υποστηρίζουν μεγάλες εταιρείες. Σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση που είχαμε με την ε, Ένωση των Βιομηχάνων από τη δική μου σκοπιά, ε, μπορώ να σας πω ήταν κάπως μυθική και πολύ ψυχρή στις παρεμβάσεις του. Θεώρησαν ότι το θέμα του ΠΟΕ είναι τελείως διαφορετικό, ότι θα μπορούσε να μείνει και εκτός ΠΟΕ και ότι η κυβέρνηση θα λάβει κάποια μέτρα για να αποφύγει τα αρνητικά, τις αρνητικές συνέπειες της ένταξης. Επίσης, ε, μας είπαν οι επιρρώσεις επιχειρηματίες ότι η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, ήταν όπως θα ήθελαν τώρα. Στην επίσκεψη στη Δούμα μας αναγνώρισαν οι βουλευτές ε, ότι, υπήρξε, ότι δεν υπήρχαν πολιτικοί λόγοι για να καταψηφίσουν αυτές τις ε, την προσχώρηση, οι περισσότεροι υπερψήφισαν για οικονομικούς λόγους. Για τι μη κυβερνητικές οργανώσεις μας είπαν ότι είναι διεφθαρμένο όλο το σύστημα στη Ρουσία, όλες οι επιχειρήσεις είναι διεφθαρμένε ή διευθύνονται και εμένα με εντυπωσίασε πραγματικά αυτό, γι' αυτό ρώτησα τον ε, εκπρόσωπο με τον οποίο συναντηθήκαμε ότι ε, πώς ε, θεωρούσε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει η δική του με κυβερνητική οργάνωση και αν υπάρχει ελπίδα. Αλλά μου είπε ότι υπάρχει, υπάρχει ελπίδα γιατί αρχίζουν τώρα να αντιλαμβάνονται οι πολίτες τη διαφθορά ως πρόβλημα. Και επίσης η επίσκεψη στο ήταν πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος ε, γιατί επισκεφθήκαμε αυτό το χώρο ε, όπου υλοποιείται έρευνα και καινοτομία. Συμπερασματικά να σας πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το ταξίδι. Εμείς μπορούσαμε να δούμε ότι η θέση της Ρωσίας στον ΠΟΕ αυτή τη στιγμή συνεχίζει να μην είναι και τόσο ξεκάθαρη και επίσης ε, οι πληροφορίες που λάβαμε θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για τις διαπραγματεύσεις, τις μελλοντικέ που θα έχουμε με τη Ρωσία. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σα Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφέρω τέσσερα σημεία τα οποία μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Αφενός, το έδειξε προηγουμένω και οι συνάδελφοι, η Ρωσία είναι βέβαια στον ΠΟΕ, αλλά από ό,τι φαίνεται η Ρωσία δεν αποδέχεται του κανόνε του ΠΟΕ. Και πιο συγκεκριμένα, έχουν νομιμοποιηθεί τα προστατευτικά μέτρα για να σταθεροποιηθεί η δική της οικονομία, κάτι που αντίκειται στους κανόνες του ΠΟΕ. Παραδείγματος χάνει ο φόρος για την ανακύκλωση. Εδώ λοιπόν ε, κατ' ουσίαν καταβάλλονται προσπάθειες, ε, ε, τα περιορισμένα έσοδα του κρατικού προπολογισμού να τα εξισώσουν με άλλους κανονισμούς, να βρουν ισοδύναμα. Ξέρουμε ότι ε, οι δασμοί είναι σημαντικό εργαλείο για τη Ρωσία για να σταθεροποιήσει τον προπολογισμό της. Αυτό όμως δεν αποτελεί δικαιολογία για να παραβιάζονται οι κανόνες του ΠΟΕ. Δεύτερον, υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα. Στη Ρωσία ε, είναι δυνατόν, εξακολουθεί να είναι δυνατόν να δορδοκίσει οποιοδήποτε. Υπάρχουν λοιπόν κανόνες Αναφέρθηκε το παράδειγμα της IKEA. Η IKEA για δύο ολόκληρα χρόνια αρνήθηκε να καταβάλει τις ε, μίζες και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούσε να ανοίξει υποκατάστημα στη Ρωσία. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό σημείο το οποίο πρέπει να αναφέρουμε. Οι ε, ισότιμες εμπορικές ανταλλαγές μπορούν να λάβουν χώρα, δίκαιο εμπόριο, μόνο εφόσον δεν υπάρχει διαφθορά. Κάτι άλλο. Ε, πρέπει να σας πω ότι θα έλεγα ότι εξοργίστηκα όταν ετέθη το θέμα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας, κυρίως στον ενεργειακό τομέα. Σε αυτόν λοιπόν τον τομέα μας είπαν ξεκάθαρα ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να είναι εταίρος της Ρωσίας, τότε θα πρέπει να συμπεριφέρεται ως τέτοιος και μας είπανε Κοιτάξτε, εμείς οι Ρώσοι είμαστε εκείνοι που θα ορίσουμε τι ακριβώς σημαίνει εταίρος. Αυτή λοιπόν η ε, διελκυστίνδα εξουσίας δεν νομίζω ότι ευνοεί μια εταιρική σχέση και μάλιστα φτάσανε μέχρι του σημείου οι προσπάθειές μας ε, να διαφοροποιηθούμε στον τομέα της ενέργειας, ε, ο αγωγός Ναμπούκο, παραδείγματος χάρη, αμφισβητήθηκε, γιατί υποτίθεται ότι ο αγωγός αυτός αντίκειται στη συνεργασία με τη Ρωσία και μας είπαν λίγο πολύ να εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο στον South Stream ή ε, στο ενεργειακό μας πακέτο, εκεί όπου υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις που θίγουν την Gazprom. Gazprom. Μας είπανε ούτε και αυτές μπορούν να περάσουν. Άρα δηλαδή κατά τους ε, Ρώσους εταιρική σχέση. Ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει να προάγονται μόνο τα συμφέροντα της Ρωσίας. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Τέταρτον, η ρωσική πλευρά δήλωσε με απόλυτη σαφήνεια ότι στο μέλλον οι εμπορικές σχέσεις δεν θα ορίζονται σε διμέρες επίπεδο, αλλά θα υπάρχει η Τελωνιακή Ένωση με τη Λευκορωσία και το Καζακστάν. Αυτό όμως είναι πρόβλημα, γιατί η Λευκορωσία και το Καζακστάν δεν θα έλεγα ότι είναι χώρος δημοκρατίας. Την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Καζακστάν. Και δεύτερον, Όλα αυτά ε, ξέρετε ε, έχουν και το ότι το αφεντικό στο που απλά σε αυτή τη σχέση είναι η Ρωσία. Άρα δηλαδή εδώ καταβάλλονται προσπάθειες ε, να μην μπει κανεί στην ουσία των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στο μέλλον. Δηλαδή να έχουμε κατά νου ότι δεν είναι δυνατόν ορισμένοι να θέλουν να επιβάλλουν τη μουσική που θα ακούν όλοι οι εταίροι. Ευχαριστούμε, Μπέντ. Επειδή δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει, να δώσω απευθεία το λόγο στην Επιτροπή, τον εκπροσωπό Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίως, συμφωνούμε με τα περισσότερα από τα μέλη που εντόπισαν συγκεκριμένα προβλήματα. Ήταν πολύ χρήσιμη επίσκεψη. Μάλλον με την αφορμή του σχολιασμού τη χρήσιμη αυτή επίσκεψη, όπου ξέρετε ότι συμμετείχαμε και εμεί μαζί με του εκπροσώπου του Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα, ω προ τον ΠΟΕ και την υλοποίηση των σχετικών διατάξεων, συμφωνούμε με τι ανησυχίε των ε, βουλευτών. Ξεκινήσαμε εντατικέ ε, διαπραγματεύσει με του Ρώσου εταίρου μας, προκειμένου να δούμε τι γίνεται με κάποια μέτρα για την ε, γεφύρωση των ε, διαφορών, όπως ας πούμε ο, φόρος, ο δασμός ανακύκλωσης για τα εισαγόμενα οχήματα. Την εισαγωγή ζών των ζώων. Εκεί βρίσκουμε ε, τα αίτια που χρησιμοποιεί η Ρωσία, οι δικαιολογίε να είναι τελείω ασταθεί από υγειονομική και φυτογειονομική άποψη. Επίση, οι συμφωνημένοι δασμοί για τα 270 για τα 370 ήδη δεν ε, εφαρμόστηκαν με κόστος πολύ μεγάλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά είναι απλώς μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχουμε λοιπόν εντατικέ διαπραγματεύσεις με τις ρωσικές αρχές επί των θεμάτων αυτών, προσπαθώντας να βρούμε λύσεις ε, χωρίς ε, να υπάρξει σύγκρουση. Όμως μπορεί να υπάρξουν και άλλου είδους λιγότερο φιλικές διευθετήσεις αυτών των ε, διαφορών λόγω της μη εφαρμογή μέτρων. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες των ε, βουλευτών για αρκετά προβλήματα όπως αυτό το φαινόμενο της διαφθοράς που όλοι το σχολίασαν. Πρέπει να πω σχετικά ότι πολλά από τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων ε, σε σχέση με τις ε, νέες μας συμφωνίες θα πρέπει να δούμε να... και τι πρόοδο θα κάνουν οι αρχές στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος, ιδίως στις δημόσιες προμήθειες. Οι ρωσικές αρχές στο ανώτατο επίπεδο έχουν οι ίδιες στήξει αρκετές φορές το φαινόμενο της διαφθοράς. Επίσης, σημειώνουμε και συμφωνούμε με αυτό που υπόθηκε για τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα ή τέλος πάντων να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους των διαπραγματεύσεων από τις διμερείς συμφωνίες σε διαπραγματεύσεις με μη μέλη του ΠΟΕ. Πράγμα που από δική μας πλευράς δεν μπορεί να θεωρηθεί εφικτό. Όπω η εμπορική συμφωνία τη Ρωσία με το Καζακστάν. Το έχουμε εξηγήσει αυτό στου Ρώσου εταίρου. Εκεί δεν υπάρχει συνέπεια. Θα πρέπει λοιπόν οι δικέ μα διαπραγματεύσει να εντατικοποιηθούν. Πιστεύουμε ότι είναι ουσιώδου σημασία αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην ξεχνάμε ότι ο πρώτο ε, εμπορικό εταίρο τη Ρωσία είμαστε εμεί. Και μακράν απέχουμε από του υπόλοιπου. Άρα. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε πολύ καλύτερη μεταχείριση για τους Ρώσους ε, στις διμερείς μας διαπραγματεύσεις από ότι για οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΠΟΕ. Εδώ θα πρέπει να δούμε και τι ενδιαφέρον θα παρουσιάσει η ρωσική οικονομία και οι σχετικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα, διότι ακούστηκαν δημόσιες δηλώσεις στη Ρωσία για το ότι πρέπει η χώρα να βρεθεί μεταξύ τις πρώτες 20 χώρες που προσελκύουν ξένες επενδύσεις, που θα πρέπει να κάνει πιο ποικίλη και ενδιαφέρουσα την οικονομική δραστηριότητα, να δει τι θα γίνει με την εξαγωγή ενέργειας και καυσίμων, να αναζητήσει ισχυρότερου εμπορικού εταίρου μέσα των διαπραγματεύσεων για τη νέα μα εμπορική συμφωνία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Θα... Δεν βλέπω να θέλουν άλλοι το λόγο. Σας ευχαριστώ, λοιπόν. Καλό θα ήταν να γνωρίζει το περιεχόμενο του ψηφίσματό μας ε, η Ρωσία, η ρωσική πλευρά. Αυτό που είχαμε στην τελευταία ολομέλεια για την ε, προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Και το τι συνέχεια δόθηκε σε αυτό με το monitoring group, με την ομάδα, τη διευθύνης ομάδα. Θα πρέπει λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με τη συνέχεια του θέματος αυτού. Θα το παρακολουθούμε στενά. Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε στο σημείο 9, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Το πρώτο σημείο, σημείο 9, είναι μεταβατικές ρυθμίσεις των πλαισιδημερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μέλων και τρίτων χωρών. Ο κανονισμό ΠΙΤ, όπω λέγεται, προθεσμία κατάθεση των υπολογιών ήταν η 9η Νοεμβρίου και δεν ε, είχαν κατατεθεί τροπολογίε. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία. Έχουμε μόνο την τελική ψηφοφορία και φυσικά πρέπει να είναι ηλεκτρονική η ψηφοφορία αυτή. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. So Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγητή που ήταν και πρόεδρος, ο πρόεδρός μας ήταν ο εισηγητής. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 10 ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότηση στι πτυχέ που αφορούν την ανάπτυξη δικαιωμάτων διανοητική διοκτησία σε θέματα γενετικών πόρων, οι επιπτώσει στη μίσο τη φτώχεια στι αναπτυσσόμενε χώρε. Ο Εισηγητή είναι ο κύριο Σόλτ και έχουμε ένα μακρύ κατάλογο ψηφοφοριών. Σα παρακαλώ να είστε όλοι συγκεντρωμένοι. Λοιπόν, να περάσουμε καταρχήν στην τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Να περάσουμε λοιπόν στη συμβασμό 2. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμό 3 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, εποχές να το ελέγξουμε. Την τροπολογία 11, άρχεται ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Να περάσουμε στην τροπολογία 13, υπέρ. Κατά. Αποχές. Και την 13 να την ελέγξουμε. Μάλιστα, ήταν σαφές. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Να περάσουμε στην τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε και αυτή. Άρχεται η ψηφορία για το 14. Πέρας. Εγκρίνεται. Να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 13 ψήφοι υπέρ, καμία κατά, 12 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 11. Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, Εφενό και τη Κολομβίας και του Περού αφετέρου. Όπω ξέρετε, είχαμε πολλέ συζητήσει για το θέμα αυτό και τώρα ήρθε ο καιρό να λάβουμε αποφάσει. Δύο ομάδε έχουν ε, καταθέσει τροπολογίε για να αρνηθούν τη συνένεση. Θέλω να σα ευχαριστήσω όλου που συμμετείχατε ενεργά σε αυτή τη συμφωνία για το ενδιαφέρον σα και θα ήθελα να καλωσορίσω και του εκπροσώπου και των δύο χωρών που είναι παρόντε εδώ στη σημερινή ψηφοφορία. Να περάσουμε τώρα στην τροπολογία υπαρτιμών 1 και στην τροπολογία 2. Είναι ταυτόσιμες. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Να περάσουμε στο σχέδιο της σύστασης, έτσι όπως δεν έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 ψηφί υπέρ, 4 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον Μάριο Δαβίδ που ήταν ο του φάκελου αυτού. Θα ήθελα τώρα να περάσω στο σημείο 11α που προσθέθηκε στην μερική διάταξή μας θα επανέλθουμε στην πρόταση Omnibus 1 για το εμπόριο που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο στις 14 Μαρτίου μετά από προπαρασκευαστική δουλειά. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν τώρα είναι έτοιμοι να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις για μια πιθανή δεύτερη ανάγνωση. Και σύμφωνα με τις γενικές αρχές ε, για τις τακτικές κανονικές διαδικασίες θα πρότεινα να λάβουμε τις εξής αποφάσεις. Καταρχήν, να μπούμε σε άτυπες διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και την Κομισιόν προκειμένου να καταλήξουμε σε μια έγκαιρη δεύτερη συμφωνία ανάγνωση. Επίσης, το ψήφισμα της 14 Μαρτίου αποτελεί στη βάση της διαπραγματευτικής ομάδας και τρίτων. Και το εκτιμώντας από το Omnibus 2 σε σχέση με την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποτελέσει μέρος των διαπραγματεύσεων και επίσης η διαπραγματευτική ομάδα θα, ε, στην διαπραγματευτική ομάδα θα συμμετέχει ο κύριος Μοηρέιρα, ο κύριος Βησαντρόβο και οι ισκιώδεις από τις άλλες ομάδες. Να περάσουμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ. Δεν υπάρχουν ε, αποχές, δεν υπάρχει καταψήφιση. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις ψηφοφορίες Σας ευχαριστώ όλους. Και θα ήθελα τώρα να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για να αποχωρήσουν οι συνάδελφοι. Dear colleagues and dear uh, ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, εάν θέλετε οι ομιλίε εκτό αίθουσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν περάσουμε στο σημείο 12, να δούμε το 12 νέο, το Α, γιατί χθε οι συντονιστέ αποφάσισαν να συμπεριλάβουν στην ημερήσια διατάξη ανταλλαγή απόψεων με τον, με τον εκπρόσωπο τη Επιτροπή για τον κανονισμό κανόνων προέλευση. Η πρόταση έγινε από την πρόεδρο μα, κυρία Μοσκαρντίνη. Όπω ξέρετε, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε με ευρία πλειοψηφία την θέση πρώτη αναγνωσή το 2010 και έκτοτε το Συμβούλιο δεν έκανε τίποτα για τον κανονισμό αυτό. Ακόμη και μετά από πολλές, ε, ε, πολλά αιτήματα του Ευρωκοινοβουλίου. Τώρα, μια εξέλιξη που μας εξέπληξε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε του χρόνου θα ανακαλέσει τον κανονισμό. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να αιτιολογήσει αυτή την ε, πρόθεσή της θα αντικαταστήσει τον κανονισμό αυτό με κάποιον νέο. Πριν δώσω βέβαια το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δώσω το λόγο στην ε, αντιπρόεδρό μας για το θέμα αυτό, την κυρία Μουσκαρντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόβλημα με τον κανονισμό αυτό είναι πρόβλημα πολιτικού χαρακτήρα και τεχνικού αλλά και θεσμικού. Το κοινοβούλιο μας τον Οκτώβριο του 2010 ψήφισε και υπερψήφισε με ευρία πλειοψηφία τον κανονισμό αυτό. Και μάλιστα επειδή βελτιώθηκε με τις τροπολογίες της δικής μας Επιτροπής και από συναδέλφους όλων των πολιτικών ομάδων. Σε εκείνη την ε, στιγμή ο κύριος Δεχούχτη είχε εκφράσει την ε, μεγάλη του εκτίμηση για, την, ε, για τον κανονισμό όπως τον ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο. Μετά όμως έχουμε δύο χρόνια σιωπή και στις 22 Οκτωβρίου φέτος ο κύριος Δεχούχτ ε, μας ενημερώνει ευνηδίως για την απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων να αποσύρουν τον κανονισμό αυτό. Και μάλιστα την επομένη ημέρα το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013 δεν περιλαμβάνει καν τον κανονισμό αυτό. Ουδέποτε όμως υπήρξε παραμικρή επικοινωνία με την Επιτροπή μας, ούτε με το Ευρωκοινοβούλιο μετά την Ολομέλεια εκείνη. Εφόσον λοιπόν μια τέτοια, ένα τέτοιο νομοθέτημα ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο στην ε, πρώτη ανάγνωση και υπήρξε και μια τόσο ισχυρή δήλωση από την πλευρά του Επιτρόπου Βεβαίω και δικαιούται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει και να ανακαλέσει ε, ένα νομοθέτημα που έχει ψηφιστεί στην πρώτη ανάγνωση, αλλά μόνον εφόσον έχει αιτιολογήσει ενώπιον του Κοινοβουλίου του λόγου τη ανάκληση αυτή. Για αυτού του λόγου, ο Επίτροπο Δεχούχτ προσφάτως ενημέρωσε το Κολέγιο των ε, Επιτρόπων, αλλά ουδέποτε φρόντισε να αιτιολογήσει την απόφαση αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό. Πρέπει να δούμε την ουσία των ε, κινήτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ τα κοίταξα και τα βρίσκω τελείως ε, ανεπαρκή. Ακόμη και η επιστολή που μου απεστάλθη από τον κύριο Ντεχούτ πριν τέσσερι μέρες που σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσε να υποκαταστήσει μια επίσημη συνάντηση με τους εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου, διότι πρόκειται για... είμαστε ένα σώμα δημοκρατικά εκλεγμένο. Πρέπει να υπερασπιστούμε τις ε, αρμοδιότητές μας. Θα ακούσω λοιπόν με ε, ιδιαίτερη προσοχή μαζί με τους συναδέλφους αυτά που θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν κάτι έχει να πει σχετικά, και έπειτα Ελπίζω να συνεχιστεί η συζήτηση και φαντάζομαι ότι και άλλοι εισηγητέ, σκιώδεις εισηγητέ για το θέμα αυτό, ο κύριος Ρινάλντι, ο κύριος Σούστα θα έχουν κάτι να πούν σχετικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, στον κύριο Παλό Καλτσότη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Αντιπρόεδρο Μουσκαντίνη που μας έκανε την εισαγωγή για το σημείο αυτό. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει καμία βιβλία για το πώς η Κομισιόν και ο Επίτροπος Δεγκούκτ σέβεται αυτό το θεσμό η πρόθεση να προτείνει στην Επιτροπή να αποσύρει αυτόν τον κανονισμό γνωστοποιήθηκε στον Πρόεδρο πριν ε, να λάβει απόφαση Κομισιόν και όπως ε, σας είπα είναι απόφαση Κομισιόν και όχι του Επιτρόπου, λεφθέντος αυτού. Είναι αλήθεια και παραμένει αληθές ότι η Κομισιόν δίνει πολύ μεγάλη σημασία στους στόχους που ήθελε να καλύψει ο κανονισμός και αναφέρομαι κυρίως στην ενημέρωση του καταναλωτή για την προέλευση των αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους η Κομισιόν αποφάσισε να αποσύρει τις προτάσεις είναι πολύ. Καταρχήν, έλαβαν υπόψη το γενικό πλαίσιο. Ένα, υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία που επισέρχονταν. Καταρχήν. Και υπό την επιφύλαξη των σημαντικών προσπαθειών της Κομισιόν να βγει από το διέξοδο, ήταν σαφές ότι η πρόταση όπως προβλεπόταν το 2005, αλλά και όπως τροποποιήθηκε από το κοινοβούλιο αυτό, δεν πρόοδευε στο Συμβούλιο, δεν σημείωνε πρόοδο στο Συμβούλιο. Επομένω, ήταν δύσκολη η κατάσταση και έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Δεύτερον, από τεχνική σκοπιά, κατά τη διάρκεια αυτών των 7 ετών, υπήρξε εξέλιξη της νομολογίας του ΠΟΕ. έτσι ώστε οι παράμετροι σύμφωνα με τις οποίες ε, ένα σύστημα σημειώση της προέλευσης θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι σέβεται πλήρως του κανόνες του ΠΟΕ, άλλαξε. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι θα σεβόμαστε το δίκαιο του ΠΟΕ, θα ήταν προτιμότερο να έχουμε μία πρόταση που να ισχύει όχι μόνο για τα εισαγόμενα προϊόντα, αλλά και για τα εγχώρια. Για αυτό το θέμα, και αυτό είναι τεχνικό ζήτημα, θα χρειαζόμασταν μια πρόταση που να μην βασίζεται στο 207 της Σύνδεξης Λειτουργίας τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στο 144. Γιατί θα είχαμε έναν κανονισμό που θα αφορούσε και την εσωτερική αγορά προκειμένου να καθορίσουμε αν χρειάζεται δράση δυνάμει του άρθρου Καταρχήν θα έπρεπε να δούμε αν υπάρχουν ε, εμπόδια στο εμπόριο λόγω αποκλήσεων και αν χρειάζεται ένα νέο σύστημα για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών. Η εξέταση αυτή μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι προκειμένου να αναλάβουμε δράση για το θέμα αυτό, πρέπει να ακολουθηθεί μια νέα οδός και όχι αυτή που είχαμε ξεκινήσει το 2005. Υπάρχουν και κάποια τεχνικά θέματα που πρέπει να εξεταστούν, θα πρέπει να υπάρχει σήμανση στα εγχώρια αγαθά, αν θα πρέπει να λέμε ότι έχουν κατασκευαστεί παρασκευαστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε κάποιο κράτος μέλος κτλ. Αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους η Κομισιόν αποφάσισε να αποσύρει την πρόταση ε, του 2005 σε ό,τι αφορά τώρα σε μια νέα πρόταση δεν ε, υπάρχει πρόθεση να υπάρξει μια πρόταση που θα βασίζεται στο εμπόριο και θα φορά μόνο σημαντικά αγαθά. Αν χρειαστεί περαιτέρω δουλειά για να επιλύσουμε τα ζητήματα αυτά από μια ευρύτερη προοπτική, δηλαδή να δούμε και την εσωτερική διάσταση, θα πρέπει φυσικά να ολοκληρωθεί η συζήτηση στην Κομισιόν καταρχήν για το θέμα αυτό μεταξύ των διάφορων ε, αρμόδιων επιτρόπων. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση η αρμόδια επιτροπή για την εσωτερική αγορά και για τις επιχειρήσεις θα το διερευνήσουν αυτό το θέμα. Όπως σας είπα, ξεκολουθούμε να επιθυμούμε την ίδια αρχή, αλλά δεν πιστεύουμε ότι τελικά ένας κανονισμός δεδομένου του πλαισίου που σας περιέγραψα, τελικά θα εξυπηρετούσε τους στόχους και τους σκοπούς καταλήλως. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ Πρόεδρε για το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριος Σούστα πρώτος και μετά η κυρία Κέλλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής που μας ενημέρωσε σε θεσμικό επίπεδο για μια απόφαση που από πολλές σκοπιές ήταν αναμενόμενη, ωστόσο μας ευνηδίασε. Απλούστερο θα ήταν εάν ο Επίτροπος Δεχούχτ είχε πει αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ότι στο Συμβούλιο ουδέποτε επετεύχθη η πλειοψηφία για να ληφθεί απόφαση για αυτό το θέμα. Και με τον καιρό και ο ίδιος ο Επίτροπος άλλαξε γνώμη. Διότι το να θεωρηθεί ή να σχολιαστεί μια πρόταση ως ε, απερχιωμένη, ως ξεπερασμένη, είναι μια προσωπική εκτίμηση. Δεν αλλάζει όμως κάτι αυτό. Αν ήταν απερχιωμένη πριν μια μέρα θα ήταν το ίδιο και πριν μισή χρόνια. Το θέμα είναι πολιτικού χαρακτήρα όμως περισσότερο και θα μπορούσε να επιληθεί εάν λαμβάναμε υπόψη τα εξή. Ότι η θεμελίωση της απόφασης αυτής με, με τους νέους κανόνες του ΠΟΕ για προϊόντα όπως ο καπνός, ο τόνος που μικρή σχέση έχουν ε, με το σήμα Made in. Εκεί έχουμε αρχές ένδειξης γεωγραφικής προέλευσης για αγροτικά και προϊόντα και τρόφιμα. Αλλά όχι τα προϊόντα αυτά που θα διευθετούσε ο κανονισμός αυτός με τις διατάξεις του. Το πρόβλημα λοιπόν θα μπορούσε να επιληθεί με απλούστατο τρόπο. Η δυσκολία όμως είναι ότι στην Ευρώπη το να επιλύουμε με απλό τρόπο τα προβλήματα δεν φαίνεται να γίνεται συχνά θα παίρναμε δύο γραμμές από την νομοθεσία των ΗΠΑ για κάτι που θεωρείται ως θέμα που ρυθμίζει το Made in USA. Κάτι που είναι υποχρεωτικό για όλους, για την αντικειτοθεσία στις ΗΠΑ, ώστε να επιλύεται το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι εάν αλήθευε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Αλλάζοντα του κανόνες μας δεσμεύει και μας υποχρεώνει να αποσύρουμε τον κανονισμό ή έστω να αλλάξουμε τελείως την προσέγγιση μας, την νομοθετική προσέγγιση στον κανονισμό, τότε θα έπρεπε να ξεκινήσουν διαδικασίες σχετικέ και για τις υπόλοιπες χώρες. Κίνα, Ηνωμένε Πολιτείε, Καναδάς, Αυστραλία, Ιαπωνία, διότι οι δικοί τους κανόνες για την ε, σήμανση των προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες θα ήταν τεχνικός φραγμός. Άρα θα παραβιάζονταν οι κανόνες του ΠΟΕ. Η νέα λοιπόν αυτή ρύθμιση του ΠΟΕ δεν θα δημιουργούσε προβλήματα, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα ή ως αιτιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάζει τους κανόνες της. Θα γινόταν ένα θέμα ε, διαφοράς και μια διαδικασία, θα ξεκινούσε μια διαδικασία επίλυσης διαφοράς ευρύτερη για όλες τις σχετικέ περιπτώσεις. Σκόπιμο νομίζω ότι είναι λοιπόν να υπάρξει συντονισμός των ε, σχετικών προδιαγραφών που αφορούν τα προϊόντα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίω να υπάρξει και ευθυγράμμιση με τα όσα ισχύουν για τα προϊόντα από τρίτε χώρες. Είναι κάτι που όλοι το επιθυμούμε. Σε λίγες ώρες θα μιλήσουμε για τους δημόσιου διαγωνισμού και τους κανόνε αμοιβαιότητα. Εδώ λοιπόν αμοιβαιότητα θα πρέπει να αναζητούμε και στους κανόνες του εσωτερικού εμπορίου. Μεταξύ μάλλον εσωτερικού εμπορίου και εξωτερικού εμπορίου. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουδέποτε θέλησε να το καταλάβει. Γιατί από καταβολή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε δεν ήθελε να καταλαβαίνει τέτοια θέματα εις βάθος. Υπάρχει ένας ε, προστατευτισμός εδώ, μεταμφιεσμένος, και η υπεράσπιση ενό απερχαιωμένου παραγωγικού συστήματο. Όλοι οι τομεί που αναφέρονται στον κανονισμό είναι τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει πάρα πολύ μεγάλε δόσει καινοτομία. Και αφορά αυτό ιδιαίτερω και του καταναλωτέ. Ε, κάνω έκκληση λοιπόν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω θεσμικό όργανο που έχει το, την αρμοδιότητα τη πρωτοβουλία, τη νομοθετικής πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά πρώτον, να σεβαστεί τα άλλα θεσμικά όργανα. Είναι τόσο ανόητο να μην έχει γίνει σεβαστό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια τέτοια περίπτωση. Έπειτα, για θέματα που προκαλούν ε, ίσως αμφιβολίες σε σχέση με τους κανονισμούς αυτού και απαιτούνται αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί το Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι απλώ ένα εξωγήινο σώμα που βλέπει τα θέματα διαφορετικά και χρησιμοποιεί αιτιολογήσει τελείω διαφορετικέ από αυτέ που έχουν οδηγήσει στι αποφάσει τη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπροσωπεί 500 εκατομμύρια πολίτε στο Ευρωκοινοβούλιο και οι βουλευτέ κάποιον εκπροσωπούν από την χώρα τους, πραγματικούς ανθρώπους. Ε, Υπάρχουν οι ομάδες πίεση, υπάρχουν οι ενδιαφερόμενοι, αλλά όλοι αυτοί θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και γι' αυτό τη δίνουν τέτοια μεγάλη βαρύτητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν με περίπου 550 ψήφους ενέκρινε αυτόν τον κανονισμό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει κανείς που μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα το γενικό συμφέρον ε, της, ε, των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων από την ψηφοφορία αυτή όπως είχε γίνει. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεσμικό όργανο και όχι με μεμονωμένη επίτροπη ή ο καθένας ξεχωριστά να μην λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις που μπορεί να παραβιάζουν το ιερό δικαίωμα των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων, πού παρασκευάστηκαν τα προϊόντα. Σκοπός είναι να ευθυγραμμίζεται ανάλογα και η ε, προσέγγιση τακτική των μεγάλων εμπορικών μας εταίρων. Εάν είχαν τέτοιου κανόνες και οι εμπορικοί εταίροι μας, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αλλιώς διαπράττει σφάλμα εναντίον των 550 εκατομμυρίων καταναλωτών η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Αυτού πλήττει εφόσον δεν εξασφαλίζει κανόνες που θα τις ε, δώσουν την ε, δυνατότητα να ανταγωνίζεται με ίσους όρους τους υπόλοιπους εμπορικούς εταίρους στην παγκόσμια αγορά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, Keller, please. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να επανέλθω στο ψήφισμα για το βαμβάκι. Αυτό είναι το επόμενο θέμα. Κοιτάξτε, θα ήθελα να μιλήσω όχι ως ποιότητα του Πρόεδρου, αλλά του μέλους ε, για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, ανεξάρτητα με το αν είναι κανείς ε, υπέρ ή κατά του ε, προγραμματιζόμενου κανονισμού ε, μπορώ να ε, καταλάβω γιατί η Κομισιόν θέλει να αποσύρει αυτό το θέμα. Εκείνο όμως το οποίο που δεν καταλαβαίνω και νομίζω ότι από αυτού συμφωνούμε όλοι μας είναι ότι το Συμβούλιο για δύο ολόκληρα χρόνια δεν κάνει απολύτως τίποτε για το θέμα αυτό. Δεν είναι δυνατόν να, υπάρχει, να έχει ξεκινήσει μια νομοθετική διαδικασία, η Κομισιόν να καταθέτει πρόταση, εμείς να ψηφίζουμε σε πρώτη ανάγνωση και το Συμβούλιο να μην κάνει τίποτα. Άρα δηλαδή θα πρέπει από κοινού με το Συμβούλιο ε, να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πρέπει να συνεχιστεί το θέμα. Και δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε αυτή την πρόταση γιατί προφανώς είναι πεπισμένη ότι είναι σωστή. Και εμείς ε, στο Κοινοβούλιο ε, είχαμε ε, με τροποποιημένη πρόταση, στην τροποποιημένη πρόταση ευρεία πλειοψηφία. Άρα δηλαδή αν ε, οι τεχνικοί λόγοι είναι το πραγματικό αίτιο, τότε γιατί το πρώτο μήνυμα που περνάει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσύρει την πρότασή της και δεν είναι το πρώτο μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει νέα πρόταση. Και το δεύτερο μήνυμα να είναι ότι αποσύρεται η πρόταση. Συγκεκριμένα δηλαδή, συγκεκριμένα ρωτώ το εξή. Η Κομισιόν ήταν πεπισμένη όταν έκανε την πρώτη πρόταση. Και τους επόμενους μήνες τι θα γίνει. Θα καταθέσει νέα πρόταση ή κατά την άποψη της Επιτροπής πάει το θέμα, έχει χαθεί τελείως. Η Κομισιόν παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχήν θέλω να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλιά σας ε, ότι πράγματι ε, δεν υπήρξε καμία κίνηση τα τελευταία δύο χρόνια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε προσπάθειες έτσι ώστε να κρατηθεί η συζήτηση στο Συμβούλιο. Όσον αφορά τώρα το ερώτημά σας σχετικά με το κατά πόσον θα κατατεθεί άλλη πρόταση ή όχι, εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ε, απαντήσω σχετικά με την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή τη φάση η Κομισιόν έχει αποσύρει την πρότασή της και δεν πιστεύει ότι η ε, πολιτική εμπορίου είναι η σωστή πολιτική Δηλαδή δεν πιστεύει ότι μέτρα που θα ληφθούν που θα επηρεάζουν μόνο τις εισαγωγές, δεν πιστεύει η Επιτροπή ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση στο πρόβλημα το οποίο έχουμε εντοπίσει ε, και το οποίο επιθυμούμε να επιλύσουμε. Και ας μην ξεχνάμε υπάρχουν ε, οι συγκεκριμένε εξελίξεις στο Συμβούλιο και στην ομολογία του ΠΟΕ που δεν ήταν η ίδια το 2009 τον Οκτώβρη όταν δηλαδή το, το Κοινοβούλιο υπερψήφισε με 525 ψήφους υπέρ αυτής της πρότασης, αν θυμάμαι καλά. Ε, τροποποιήθηκε αυτή η απόφαση και Δυστυχώς η νομολογία του ΠΟΕ ισχύει και για τα βιομηχανικά και τα αγροτικά προϊόντα. Ο τόνος ε, δεν θεωρείται ούτε βιομηχανικό ούτε αγροτικό προϊόν. Σε αυτή τη φάση λοιπόν υπάρχει το εξής ε, σαφές μήνυμα από τον κύριο Σούστα και από ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου να αναλυφθεί η δράση, να ξεκινήσει ο κανονικός διάλογος ανάμεσα στους ε, θεσμούς. Όπως είπα ήδη λοιπόν, αν έπρεπε να κάνουμε κάτι ανάλογα με αυτά που υπάρχουν τώρα, πιστεύουμε θα έπρεπε να δραστηριοποιηθούμε στο θέμα ε, των εισαγωγών και όχι ε, να αναλυφθούν μέτρα ε, βιομηχανικής πολιτικής. Ε, δεν νομίζω ότι μπορώ να σας πω τίποτα άλλο από αυτού αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Μουσκαρντίνη. Κοιτάξτε, λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκαστήκατε να έρθετε εδώ σε μας και να μας πείτε ανοησίες. Διότι αν ο κανονισμός του ΠΟΕ τροποποιήθηκε το 2009, αυτό σημαίνει ότι ο Επίτροπος Δεγκούτε δεν έχει πλέον αρμοδιότητες και αυτός ο αναρμόδιος ήρθε εδώ και μας έφερε ένα κανονισμό που πρέπει να τροποποιηθεί και ποτέ επ' αυτού ψηφίσαμε. Εάν λοιπόν αυτά ψηφίσαμε τα 2010 μετά την τροποποίηση των κανόνων του ΠΟΕ και ακόμα ε, ένα χρόνο αργότερα ψηφίσαμε πάλι για κάτι που δεν υπήρχε ή εσείς ε, στην Κομισιόν ε, κοιμόσασταν ή ε, δεν ήσασταν καθαροί. Δεν θέλω να απαντήσετε τώρα γιατί κοιτάξτε, εδώ εμείς θέλουμε τον θεσμικό σεβασμό και δεν μπορείτε να μας κοροϊδεύετε. Μπορεί ε, κανείς ε, πολιτικά να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν είναι δυνατόν να εξευτελίζει το Κοινοβούλιο και να γράφει γελία πράγματα. Μάλιστα, στην ε, επιστολή που στείλατε σε μένα στην εισηγήτρια λέτε ότι κανείς από το Συμβούλιο δεν ζήτησε να προχωρήσει αυτός ο κανονισμός ότι το Κοινοβούλιο δεν ποτίθεται κινητοποιήθηκε. Αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτά. Εσείς πότε ανακαλύψατε ότι είναι σημαντικό να εστιαστεί η εξωτερική αγορά με την εσωτερική αγορά. Κοιτάξτε, εγώ όταν αγοράζω ένα πράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, δεν μου χρειάζεται να ξέρω πού κατασκευάστηκε, γιατί κατασκευάστηκε με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Εκείνο όμως που κατασκευαστηκε γιατι κατασκευαστηκε με βαση τους ευρωπαικους κανονισμους εκεινο ομω που πρεπει να ξέρω είναι όταν έρχονται προϊόντα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί δεν υπάρχει σιγουριά ότι έχουν εφαρμοστεί οι σωστοί κανόνες. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτό, ας μην συζητάμε από αυτό. Εγώ ε, ερωτώ, πρώτον, η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι άλλαξαν οι κανόνες του ΠΟΕ. Δεύτερον, ερωτώ, τον προηγούμενο μόλις μήνα ανακάλυψε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και για κανόνες για την κοινή αγορά και όχι για την εξωτερική διεθνή αγορά. Τρίτον, για ποιον ακριβώς λόγο η Κομισιόν που υποτίθεται ότι προστατεύει τους ε, καταναλωτές βρίσκεται μπροστά σε μία τροποποίηση της νομολογίας του ΠΟΕ και δεν λέει στον ΠΟΕ να ζητήσει από τις χώρες οι οποίες ε, εφαρμόζουν κανόνες που κατά άποψή μου είναι η άποψή μα απαγορευμένες, γιατί ο δεν λέει στις χώρες αυτές να τροποποιήσουν αυτούς τους κανόνες τους. Συγγνώμη, γιατί η Κίνα να πρέπει να προστατεύει τους καταναλωτές τη και όχι η Ευρώπη. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απευθύνεται στον ΠΟΕ ε, και ε, να κοινοποιήσει ο ΠΟΕ ε, στις χώρες της αρμόδιες ότι πρέπει να τροποποιήσει τους κανόνες τους. Κοιτάξτε, ή υπάρχουν κάποια συμφέροντα ή υπάρχει κάτι άλλο. Και επ' αυτού λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά το κοινοβούλιο δεν θα ενδώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ε, παρατηρήσεις σας. Νομίζω ότι είναι ε, πολύ δύσκολο να κλείσει το θέμα αυτό αλλά εν πάση περιπτώσει ε, νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε σε μία από τις επόμενες αντίσεις μας να καλέσουμε τον Επίτροπο Ντεκούχτα να μιλήσει και για άλλα και για αυτό το θέμα και ίσως ε, πρέπει να ε, μας δώσει ο Επίτροπος πιο πολλές λεπτομέρειες, περισσότερο πολιτικές λεπτομέρειες από αυτές που έδωσε ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Εμπόριου. Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι εδώ υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Ίσως θα Μιλήσω και εγώ Ιταλικά για να είμαστε. Κοιτάξτε, η τροπολογία του νομολογία ε, του ε, ΠΟΕ έγινε το 2010 και το 2011 λοιπόν επιβεβαιώθηκε αυτή η αλλαγή της νομολογίας που σημαίνει ότι όταν εσείς αποψηφίσατε τον Οκτώβριο του 10 τότε δεν γνωρίζαμε ε, την απόφαση του εφετείων θέλετε πάνω στη συγκεκριμένη αυτή αλλαγή στον ΠΟΕ. Αυτά. Όσον αφορά τώρα στην προστασία του καταναλωτή, ο κανονισμός έχει ως στόχο να ενημερώνει τον καταναλωτή για την προέλευση, την ποιότητα, ε, όμως για αυτήν είναι αρμόδιοι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και άλλοι κανονισμοί. Μόνο η προέλευση είναι υποχρέωση. Και η Κομισιόν ποτέ δεν είπε ότι ένα προϊόν που εισάγεται από την Κίνα ή από άλλες χώρες ότι το προϊόν αυτό εξορισμού ε, δεν συμβαδίζει με την κοινοτική ε, με τους κοινωνικούς κανονισμούς. Γι' αυτό και υπάρχουν και άλλοι κανόνες. Θέλω πάντως να διευκρινίσω ότι η αλλαγή της νομολογίας του ΠΟΕ είναι μεταγενέστερη της δικής σας απόφασης και θα έχω την τιμή να εξηγήσω στην κυρία Μουσκαρντίνη ότι η αλλαγή αυτή σας λέω έγινε μετά την ψηφοφορία που έλαβε χώρα στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν έχουν αντιρρήσει συνάδελφοι, θα ήθελα να κλείσω ω εξή Υπήρξε πρόταση Κομισιόν το 2010. Ήταν πεπισμένη η Κομισιόν ότι πρέπει κάτι να ρυθμίσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2005, συγχωρείτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε την πρώτη για το θέμα αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν καλό σε μια επόμενη συνεδρίαση να συζητήσουμε με τον αρμόδιο επίτροπο για το τι θα κάνουμε με αυτό το φάκελο. Γιατί η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν δύο χρόνια αποφάσισε ότι θέλει κάτι προ αυτήν την κατεύθυνση και η Κομισιόν είχε κάνει μια πρόταση. Και νομίζω λοιπόν ότι από τη δική μα σκοπιά δεν θέλουμε μόνο απλώ ε, να μα στείλετε ένα μήνυμα ότι αποσύρεται η συμφωνία, αλλά θέλουμε να δούμε και πώ ε, θα συνεχίσουμε και τι θα κάνουμε με το περιεχόμενο. Σα ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, για τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανοιχτή του στάση. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, να περάσουμε τώρα στο σημείο 12. Τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο τη αλυσίδα ε, αξία του Μαμπακιού και θα πρέπει να συζητήσουμε το σχέδιο πρόταση ψηφίσματο για τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο τη Παγκοσμία αλυσίδα Αξία ε, του ΒΑΒΑΚΑ. Μπορεί να ε, ενταχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ε, Διεθνές Συμβούλιο και επίσης θα πρέπει να καταρτιστούν οι τρόποι να ενταχθεί στη Συμβουλευτική Επιτροπή για το Βαμβάκι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να εκφραστούν οι θέσεις μας σε σχέση με διάφορες προκλήσεις στην παγκόσμια αλυσίδα αξία του Βάμβακα. Έχουμε τι επιδοτήσει, τι ε, ασταθείς τιμέ, ε, αλλά και άλλα θέματα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, όπως είναι τα περιβαλλοντικά ζητήματα και η εξάλληψη παιδική εργασία. Το σχέδιο που ε, έχει προετοιμάσει, το έχει προετοιμάσει η κυρία Μουσκαρδίνη με την συνεισφορά του κύριου Κούντας και καλή για αυξαμένη διαφάνεια στην κοσμική λυσίδα αξίας του Βάμβακα. Και χωρί περαιτέρω χρονοτριβή, να δώσω το λόγο στην κυρία Μουσκαρδίνη. Ευχαριστώ. Όπω γνωρίζουν οι συνάδελφοι, το Βαμβάκι ε, έχει μια ένωση που λέγεται ΙΚΑΚ, όπου συμμετέχουν όλε οι κύριε παραγωγικέ χώρε. Η Κίνα, η Ινδία και οι ΗΠΑ είναι οι κυρίε χώρε παραγωγή ε, και ε, δίνει εργασία, δίνει δουλειά σε 100 εκατομμύρια οικογένειε Το βαμβάκι όμως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που έχει ένα μικρό ρόλο, παράγει το 1% της ε, παγκόσμιας ε, παραγωγής. Έχουμε 100.000 παραγωγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΙΚΑΚ. Είναι μια σημαντική ένωση, είναι ένας διεθνής οργανισμός που θα έπρεπε να εποπτεύει όχι μόνο την ποιότητα του προϊόντος, αλλά και τον τρόπο καλλιέργειας για την καλλιέργεια του βαμβακιού χρειάζεται πάρα πολύ νερό και αυτό είναι ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την χρήση γλυκού νερού αλλά και με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Όπως γνωρίζουμε εμείς στην Επιτροπή μας, το βαμβάκι είναι ένα είδος καλλιέργειας που ε, δυστυχώς, όπου δυστυχώς απασχολούνται πάρα πολύ ανήλικοι. Έχουμε εκατομμύρια παιδιά σε διάφορα σημεία του που εργάζονται στη γεωργία και συγκεκριμένα στον τομέα του βαμβακιού. Γι' αυτό ε, η δική μας ε, είσοδος στον ΙΚΑΚ, μέχρι τώρα δεν συμμετείχαμε εμείς στην Επιτροπή αυτή, αλλά συμμετείχαν ορισμένα κράτη-μέλη μεμονωμένα συμμετοχή μας λοιπόν στο ΙΚΑΚ, στην Επιτροπή αυτή, θα έπρεπε να χρησιμεύσει όχι μόνο για να προστατεύσουμε τα δικά μας συμφέροντα στον τομέα αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να υψώσουμε και μια μεγαλύτερη φωνή για το σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων και το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών στις χώρες όπου δεν έχουν γίνει σεβαστά τα δικαιώματα αυτά μέχρι σήμερα. Και Επίσης, ε, καλό ε, να ενταχθούν, ε, να καλέσουμε να ενταχθούν και άλλες χώρες όπως η Κίνα, η οποία αν και είναι η μεγαλύτερη παραγωγική χώρα, σήμερα δεν ανήκει στην ΙΚΑΚ. Γιατί δεν θέλει να σεβαστεί ούτε τους ελάχιστους κανόνες. Το πρόβλημα που είχαμε εμείς είναι το στο ιστορικό της ΙΚΑΚ ε, ψηφιζόταν, ε, ε, υπήρχε και κατά κεφαλή και εμεί ως Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύαμε να χάσουμε τις ψήφου των κρατών μελών για μία και μόνο ψήφο. Όμω τώρα, επειδή έχουμε σταθμισμένη ψηφορία, μα δίνει τη δυνατότητα να μπούμε σε αυτόν τον οργανισμό, έχοντα και την απαραίτητη επιρροή. Και φυσικά εμεί, ο ψήφισμα αυτό, ζητάμε και από την Κομισιόν να παρακολουθεί και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για το τι θα συμβεί στα επόμενα έτη μετά την είσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΚΑΚ. Και εγώ γενικά θα έλεγα ότι σας ε, παρουσίασα συνολικά το πρόβλημα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις από τους συναδέλφους, ευχαριστώ να απαντήσω. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι με αφορά, εγώ είμαι έτοιμη και περιμένω τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις και τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτή την πολύ καλή εισαγωγή στο όλο θέμα. Να δώσω απευθείας το λόγο στους συναδέλφους, ο κύριος Κούτας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω την κυρία Μουσκαρντίνη για την άριστη συνεργασία που είχαμε για το θέμα. Συμφώνησε να καλύψει και τις δικές μου μέρημνες για την παιδική εργασία και την παραποίηση προϊόντων. Να δώσω κάποιες στατιστικές βάσει του της νομοθεσίας μας υπάρχουν 250 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίω που εργάζονται σε δραστηριότητες και δράσεις και οι οποίες θα πρέπει να εξαλειφθούν. 150 εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά είναι κάτω από τα 15 και άλλα 100.000 παιδιά εργάζονται σε επικίνδυνες ε, ε, δραστηριότητες. 60% ε, εργάζονται σε αγροτικές περιοχές. Διαφορετικές μορφές παιδικής εργασίας αφορούν τις ε, χώρες που είναι παραγωγή βάμβακος παγκοσμίω και επίσης ε, στον εκοκισμό και την σπορά. Η παιδική εργασία στο γεωργικό τομέα βεβαίως δεν μπορεί να εξεταστεί άσχετα από τα πραγματικότερα αίτια, τα βαθύτερα αίτια, την ένδια και την ε, ανάγκη πρόσθετου εισοδήματο από τη νέα από τις μικρές ηλικίε, αλλά και την ελληπή προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει στα βασικά της όργανα για την εμπορική πολιτική της να απαιτεί να γίνονται σεβαστές σε όλες τις προδιαγραφές για τις εμπορικές ε, συναλλαγές. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάζει αν κατά συστηματικό ε, τρόπο μια χώρα με την οποία έχει εμπορικέ ε, σχέσεις έχει παραβιάσει τις αποφάσεις του ILO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασία, όπω την απόφαση 138 ή την 182 για την ε, απάλληψη λόγω χάρη τη παιδική εργασία σε πολλέ ε, εμπορικέ πτυχέ. Θα πρέπει λοιπόν να μα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θα λάβει υπόψη τι μέρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα τη παιδική εργασία στην τομέα τη παραγωγή Μπάμπακα και αν σκοπεύει να υποβάλει στο Ευρωκοινοβούλιο μια νομοθετική πρόταση για να προτείνει μηχανισμούς ε, εξέτασης, πραγματικής εξέτασης και αποτίμησης του κατά τα προϊόντα που παράγονται, παράγονται χωρίς την ε, παιδική εργασία. Ευχαριστούμε κύριε Κούτας. Η συνάδελφος Κέρι. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε και στο προηγούμενο θέμα και γι' αυτό συμφωνούμε και θέλω απλά να σας πω ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου εμείς ενδέχεται να καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες. Επιθυμούμε να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες γιατί θεωρούμε ότι ε, εφόσον θέλουμε να καταδείξουμε τη λύση, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταθέσουμε και συγκεκριμένες συστάσεις. Παραδείγματος χάρη, οι παράγραφοι 8 και 9. Νομίζω ότι εκεί μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, με συγκεκριμένες προτάσεις. Ε, βεβαίως, ε, αυτό δεν σημαίνει ότι διαφωνούμε, απλά επιθυμούμε να υπάρχουν πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Ένα θέμα λοιπόν, το οποίο κατά την άποψή μου είναι θετικό είναι ότι στην παράγραφο 1 Εκεί γίνεται λόγος για τη βελτίωση της διαφάνειας ε, ε, στα παράγωγα, στις αγορές ε, παραγόγων αγαθών και λίγο πιο κάτω λέτε ότι στηρίζετε τις ε, ενισχύσεις ε, στους ε, παραγωγούς βάμπακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως είναι αντιφατικό. Από τη μια λέτε ναι να χορηγούνται οι επιδοτήσεις και από την άλλη θέλετε να καταπολεμήσετε τα μέτρα στρέβλωσης του εμπορίου. Πώς το βλέπετε τελικά, τι θα επιλέξετε μεταξύ των δύο, γιατί δεν γίνεται και τα δύο ή το ένα ή το άλλο. Επίσης, ένα άλλο θέμα όπου δεν συμφωνούμε είναι εκεί που λέτε ε, σχετικά με τις απαγορεύσεις εξαγωγών και τις, ε, τους περιορισμούς. Ε, αυτή, αυτό είναι το βασικό αίτιο για τις διακυμάνσεις τιμών στο βαμβάκι. Παρότι λοιπόν συμφωνούμε ότι αυτό οπωσδήποτε παίζει ρόλο στο να καθορίζονται οι παγκόσμιες τιμές, οι τιμές βαμβακά σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει ένας πιο σημαντικός παράγον. Δηλαδή το βασικό αίτιο για την διακύμανση των τιμών του βαμβακα είναι οι αντίξωες καιρικέ συνθήκες που προκύπτουν κατά καιρούς. Και γι' αυτό το λόγο ο κλάδος αυτός ε, προσελκύει την κερδοσκοπία και όχι άλλος λόγος, ως εκ τούτου τα εθνικά συμβούλια που ρυθμίζουν την ποιότητα και την ποσότητα αυτά τα συμβούλια μπορούν ίσως να επιφέρουν τη σταθερότητα. Είτε συμφωνείτε είτε όχι, πάντως ε, οι ρυθμίσεις αυτές ε, θα επιφέρουν σταθερότητα και ε, δεν θα ρυθμίσουν τις διακυμάνσεις. Οι διακυμάνσεις έρχονται, υπάρχουν για άλλους λόγους που σας είπα. Εμείς λοιπόν ενδέχεται να καταθέσουμε τροπολογίες που θα διευκρινίζουν την κατάσταση επί της ουσίας εκείνο που θέλουν να μάθουν είναι Τι θέλετε, θέλετε μέτρα που να ε, καταπολεμούν τις τρέβλες του ανταγωνισμού ή θέλετε να συνεχίσετε να χορηγείτε ενισχύσεις στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την έκθεση που είναι περιεκτική και εξετάζει αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την καλλιέργεια βάμβακα ε, την εκμετάλλευση των εργαζομένων, κυρίως ε, το θέμα της ε, παιδικής ηλικίας. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να περιλάβουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τα φυτοφάρμακα και εκεί αναφέρεται ότι περίπου το 10% των φυτοφαρμάκων χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια του, του βάμβακα και 25% των ζανιοκτώνων επίσης. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν τις επιπτώσεις ε, και γενικότερα σε αυτούς ε, που εργάζονται στον κλάδο, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους υπόλοιπους εργαζόμενους. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κατόπιν, η χρήση του νερού και εκεί είναι ένα θέμα γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα. Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα του κόσμου είναι το ότι συρρυκνώνονται η θάλασσα στο Ουσμπεκιστάν, στα Ράλια. Άρα δηλαδή ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό παίζει ρόλο και ίσως ε, θα πρέπει να αναφέρουμε κάτι κατόπιν διαρωτώμε και κατά πόσον μπορούμε να έχουμε μια ειδική αναφορά στο Ουσμπεκιστάν. Το Ουσμπεκιστάν είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγός ε, βάμβακα στον κόσμο και έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο κατά το παρελθόν, τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ίσως θα μπορούσαμε για αυτό το λόγο να έχουμε μία συγκεκριμένη παράγραφο, ε, γιατί εγώ από ό,τι γνωρίζω θα γίνει λόγος για τα παιδιά, αλλά και για περισσότερο ηλικιωμένους, τους οποίους στο Ουσμπεκιστάν τους τελευταίους μήνες τους σέρνουν στη δουλειά. Τρίτον, συμφωνώ με αυτό που γίνεται λόγος, προβάλλεται η παιδική και η ξαναγκαστική εργασία αλλά ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο γενικοί σχετικά με τις ε, συνθήκες εργασίας σε όλους όσοι εργάζονται στον τομέα ε, συνδικαλιστικά δικαιώματα, συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και τέλος, ίσως καταθέσουμε μία τροπολογία σχετικά με την σύνθεση της Ένωσης του ΒΑΜΠΑΚΑ, του ICAC. Ίσως ε, ε, θα πρέπει και τα συνδικάτα να συμμετέχουν και αυτά για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος, ε, εξέταση περιπτώσεων κατάχρησης και το καθεξής. Ευχαριστούμε κύριε Μερφή. Δεν βλέπω άλλοι βουλευτές να θέλουν το λόγο, οπότε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της, κυρία... της Γενικής Διεθνής ΔΕΦΚΟ, τον κύριο Κίης. Ευχαριστώ. Θα σταθώ σε όλα τα σημεία, εκτός συγκεκριμένων εμπορικών πτυχών που θα, που, θα ήθελε ίσω να με συμπληρώσει ο συναδελφό μου. Ευχαριστώ την κυρία Μουσκαντίνη για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε λίγο πολύ με το σύνολο του περιεχομένου. Ευχαριστούμε και τους βουλευτές για τα σχόλιά τους, ιδίως για τα περιβαλλοντικά και τα θέματα της παιδικής εργασίας και αυτά είναι ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω χρήσιμο θα ήταν να γίνει μια σύντομη διευκρίνηση του πού βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις για να αποφευχθεί κάθε σύγχυση. Συζητούμε την προσχώρηση στην ΆΙΚΑΚ εδώ και κάποιο καιρό. Έγιναν αρκετέ συναντήσει στην ομάδα του Συμβουλίου και ουδέποτε υπήρξε απροθυμία να προσχωρήσουμε στον ΆΕΚΑ. Τα κράτη-μέλη πάντοτε έλεγαν ότι είναι υπέρ μια τέτοια εξέλιξη. Ωστόσο, η προσχώρωση ακόμα δεν είναι πραγματική, διότι είναι μακρέ οι συζητήσεις για το πώ ακριβώς θα προσχωρήσουμε. Την, στην τελευταία συνάντηση, τα κράτη-μέλη τοποθετήθηκαν λίγο πολύ ω. εξή αρχικά η συζήτηση ήταν να θα προσχωρήσουμε, όπως είπε η κυρία Μοσκαρντίνη, με κάποιο σταθμισμένο σύστημα. Ή με σταθμισμένο σύστημα να ελπίζουμε να έχουμε περισσότερες ψήφους ή με μία και μόνο ψήφο σε νέο μέλος. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν στην άποψη ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και με προσώπους της του ΆΙΚΑΚ για το να είμαστε ένα μέλος με μία συμμετοχή γενιά και μία ψήφο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ανέλαβε να το συζητήσει αυτό με τον ΆΙΚΑΚ σε άτυπο επίπεδο και με σκοπό να επιτευχθεί προσχώρηση στο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμβούν τα εξή. Ότι θα πρέπει να δει και του δικού του κανονισμού ο ΆΙΚΑΚ, γιατί αυτή τη στιγμή αποτελείται από χώρες. Δεν προβλέπεται δυνατότητα προσχώρησης μέλους, ε, οργανισμού μάλλον ως μέλους, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μπορεί να μην αποτελέσει τελικός πρόβλημα, θα μπορούσε να επιλήθει αρκετά σύντομα αυτό το θέμα. Επίσης, ως ενίο μέλος του ICAC και όπως σαφώς είπε και η κυρία Μουσκαρντίνη, θα έχουμε περισσότερη βαρύτητα θα εκπροσωπούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με αποκλειστική αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά. Θα μιλάμε λοιπόν ω ε, ενιαίο σώμα εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα όπω το περιβάλλον, η παιδική εργασία, εμπορικέ πτυχέ. Είναι ζητήματα στα οποία θα μπορούμε να επηρεάσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα. Από την άποψη του προγράμματο τώρα, λίγο δύσκολο να προβλέψουμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε ότι τώρα θα γίνουν αρκετά γρήγορα ίσω μέχρι και την επόμενη ομέλεια να μπορούμε να εγκρίνουμε τότε την ε, προσχώρησή μα, αλλά ίσω επισήμω να μην έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ελπίζουμε να γνωρίζουμε τι λεπτομέρειε τη συμμετοχή νωρίτερα και είναι και κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε και με τη Γραμματεία για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι έτοιμα. Η διαδικασία λοιπόν έχει ω εξή. Πρώτον, ο ΆΙΚΑΚ θα πρέπει να αλλάξει του κανόνε συμμετοχή Αυτό θα πρέπει να τα δουν ε, και τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό θα είναι σύντομο διαδικασία πιστεύουμε, γιατί είναι μικρές οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν. Επίτε θα πρέπει να δούμε ότι τα μέλη του ΆΙΚΑΚ δέχονται η Ευρωπαϊκή Ένωση να, συμμετέ... να συμμετάσχει ως νέο μέλος. Πράγμα που θα σημάνει και μια σχετική μείωση του προπολογισμού του ICAC, που ούτως ή άλλως δεν είναι μεγάλος. Αλλά αν δεχτεί ΆΕΚΑΚ και αποφασίσει να λειτουργεί με ένα λίγο πιο περιορισμένο προπολογισμό. Θα δούμε τι θα γίνει ή αν θα ζητήσει μεγαλύτερε συνεισφορέ από τα κράτη-μέλη του. Στην πραγματικότητα, ο ΆΕΚΑΚ έχει συγκεκριμένε συνεισφορέ από τα μέλη του. Οι δαπάνε μοιράζονται μεταξύ των μελών. Ίσως λοιπόν ε, οι επιπτώσεις από την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι και ελάχιστε όπως ο περιορισμός Στι αμοιβέ ε, του προσωπικού ή κάποιο περιορισμό κάποιων επισκέψεων. Θα δούμε πάντω ε, σε ποια νούμερα θα φτάσει ο προπολογισμό. Έτσι έχει κατάσταση ω σήμερα και ω εκπρόσωπο τη Επιτροπή, επιφορτισμένο με το θέμα αυτό, μου ζητήθηκε να το συζητήσω εγώ με του εκπρόσωπου του ΆΙΚΑΚ. Για να δω ακριβώ πού θα φτάσουν τα πράγματα. Πώ θα εξελιχθούν. Θα το συζητήσω λοιπόν με εκπροσώπου του ΑΕΚΑΚ, με τα βασικότερα μέλη, εισαγωγού και παραγωγού ε, βάμβακα για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προσχωρήσουμε στο δυνατόν συντομότερα. Thank you, Chair. Um, my name is Merloni. I'm... Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εργάζομαι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και σημειώνουμε τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου για την παιδική εργασία και εμείς τις, καταλαβαίνουμε αυτές τις ανησυχίες. Και βλέπουμε και το σημείο 7 στο ψήφισμα. Προσπάθειες για εξάλληψη της παιδικής εργασίας. Με ένα συντονισμένο και σφαιρικό πλαίσιο. Κατά την άποψή μας, ναι, αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο. Ως προς την εχνηλασιμότητα, όπως το μουσάνει τους μηχανισμούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με τις δυνατότητες να εντοπίζεται, να υπάρχει ένας ίδιος μηχανισμός εχνηλασιμότητας. Όμως η πρακτική η πρακτική δυνατότητα για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να εξεταστεί από την άποψη του κατά πόσον όλα αυτά είναι συμβατά με τον ΠΟΕ, κατά πόσον μπορεί να υλοποιηθούν και υπάρχουν και κάποια τεχνικά ζητήματα. Το κατά πόσον ο μηχανισμός αυτός δηλαδή μπορεί να είναι αποτελεσματικός όταν αφορά ένα μικρό αριθμό προϊόντων και αγαθών. Για την ώρα αυτή διεξάγουμε την, για την ώρα διεξάγουμε την σχετική ανάλυση. Περιμένουμε να δούμε και τι άλλες πρωτοβουλίες θα υπάρξουν, όπως για τον ιδιωτικό τομέα από άλλους ε, διεθνείς οργανισμούς. Σημειώνουμε πάντως το πόσο σημαντικό είναι για το Ευρωκοινοβούλιο το όλο ζήτημα. Και ένα τελικό σχέδιο, σχόλιο για τα μέτρα που μπορεί να στρεβλώνουν το εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει πολύ περιορισμένο ρόλο στον παγκόσμια στην παγκόσμια αγορά βάμβακα. Μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα του βάμβακα είχαμε το 2006 το εμπορικό σύστημα με τις επιδοτήσεις σιγά σιγά περιορίστηκε. Ειδικά για τις επιδοτήσεις που ήταν στρεβλωτικές για το εμπόριο. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία συνέπεια μεταξύ της επιδίωξης της ε, τα μείωση των στρεβλωτικών επιδοτήσεων, όπως η απαγόρευση των εξαγωγών, και το τι επιδιώκουμε σε διεθνέ επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες παρεμβάσει. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μουσκαρντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο που θα ήθελα να προτείνω εκ νέου με την ε, Κομισιόν ε, που ευχαριστώ που τοποθετήθηκε θετικά απέναντι στο κοινό μας έργο είναι ότι από τη δική μας ε, σκοπιά η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΚΑΚ θα πρέπει να επικυρώνει τη δυνατότητα για την Ευρώπη είτε να προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα είτε να προτείνει στο ιστορικό της ΕΚΑΚ τρόπους βελτίωσης της καταπολέμησης της παιδικής εργασίας και βελτίωση των περιβαλλοντικών εγγύησεων. Αν εμείς μπούμε με μια σταθμισμένη ψήφο ε, και βάσει της ε, ισχύω μας ε, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι δικές μας προτάσεις. Κατά την άποψή μου αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αλλά αν μπαίναμε μόνο ε, για να έχουμε μία ψήφο και ενώ σήμερα έχουμε 7, καθώς συμμετέχουν 7 κράτη-μέλη, εγώ νομίζω ότι δεν θα ήταν και τόσο ενδιαφέρον αυτό. Αν ε, ποτέ δεν μπορούμε ε, να ασκήσουμε την επιρροή μας. Επομένως, ήθελα να είναι σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διαθέσιμο, είναι υπέρ της ένταξής μας στην ΙΚΑΚ, αλλά με συγκεκριμένε ρήτρε που να μας επιτρέπουν ε, στο ιστορικό αυτού του οργανισμού να ασκήσουμε την ειδική μας ισχύ. Να έχουμε ένα ειδικό βάρος, όχι να έχουμε το βάρος μιας και μόνης χώρας. Τώρα, για όσα είπε οι συναδελφή θέλω ευχαριστήσω τον κύριο Κούτα ε, γιατί η συνεργασία μας για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας ε, ήταν πολύ καλή και νομίζω ότι καταλήξαμε και στα επιθυμητά αποτελέσματα. Όμως, προφανές, και αυτό το λέω σε όλους όσους έλαβαν το λόγο, εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι αν υπάρξουν τροπολογίες προς την κατευθύνση βελτίωσης της δικής μας πρότασης. και να πω ότι συνεργάστηκα με πιο στενα... από ότι με κάποιους άλλους επειδή επέδειξαν κάποιο συγκεκριμένο ενδιαφέρον για το ζήτημα. Όμως όλα όσα μπορούν να βοηθήσουν για να καταστήσουν καλύτερο αυτό το κείμενο ευχαρίστως να τα αξιολογήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά τώρα τη στρέβλωση της αγοράς. Εδώ θα ήθελα να παραθέσω το Βολτέρ και έλεγε αν θες να μιλήσεις μαζί μου θέσε τους όρους σου. Η στρέβλωση της αγοράς δεν έχει να κάνει με ενδεχόμενε επιδοτήσει στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σύστημα για ένα συγκεκριμένο είδο καλλιέργεια όπως είναι το βαμβάκι. Στρέβλωση τη αγορά, στην οποία αναφερόμαστε και είναι αυτονόητο, είναι προφανής ε, αν σε μια χώρα δουλεύουν παιδιά 8-10 ετών και αν εργάζονται άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν εισφορές, αν υπάρχουν χώρες όπου υπάρχει εκμετάλλευση της εργασίας, είναι σαφές ότι έχουμε στρέβλωση της αγοράς. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για το ηθικό ζήτημα, για την ηθισκοπιά, μιλάμε και για στρέβλωση της αγοράς. Αν μια χώρα. Τώρα αυτό δεν έχει να κάνει με το βαμβάκι γιατί είναι δύσκολο, αλλά αν πουλά στο εσωτερικό της μια χώρα και αυτό το είδαμε για τα κινέζικα φωτοβολταϊκά, ε, πουλά στην επικρατειά τη λοιπόν η χώρα αυτή σε μεγαλύτερη τιμή ένα προϊόν από ότι το πουλά στο εξωτερικό, τότε αυτό είναι dumping αν ε, απασχολούνται άτομα χωρίς να πληρώνονται, ουσιαστικά μιλάμε για στρέβλωση της αγοράς. Αν λοιπόν μια χώρα θέλει ξεκάθαρα να υποστηρίξει ένα κλάδο γιατί το χρειάζεται, αυτό είναι το ένα. Αλλά όταν εκμεταλλεύεται μια χώρα τον ίδιο της τον πληθυσμό και συνεπώς ε, θέτει στην αγορά ένα προϊόν, ε, σε ένα προϊόν, ένα προϊόν με πολύ ανταγωνιστική τιμή, τότε μιλάμε για στρέβλωση της αγοράς. Έτσι λοιπόν, σας επαναλαμβάνω, θα δεχτώ όλες τις τροπολογίες που θα αποσαφηνίσουν και θα βελτιώσουν το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής και φυσικά θα τις αξιολογήσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες στο κατάλληλο βήμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, καρποφόρο συζήτηση, επικοινωνική συζήτηση, να υπενθυμίσω σε όλου, όσοι είναι πεπισμένοι ότι μπορούν ε, να βελτιώσουν το κείμενο με τροπολογίε να τις καταθέσετε μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου στι 6 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα λοιπόν στα σημεία 13 και 14. Εκεί προβλέπεται η συζήτηση της ε, έκθεσης πρωτοβουλία της κυρίας ε, Σάιφη, όπου γίνεται λόγος για το εμπόριο και την ανάπτυξη βασισμένη στις επενδύσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και εδώ έχουμε την ε, ανακοίνωση κομισιών για το εμπόριο η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, ασχολείται με το ίδιο θέμα μέσω της πρόθεσης της ανάπτυξης μέσω του εμπορίου. Έχουμε ε, λοιπόν ε, και αμοιβέ γνωμοδοτήσεις της μίας Επιτροπής για την άλλη υπάρχουν επικαλύψει. είναι δύσκολο να έχουμε διαχωριστικές γραμμές και υπάρχουν επικαλύψεις στις δύο εκθέσει. Θα ήθελα να σε επισημάνω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στα δύο έγγραφα, τα οποία θα ψηφιστούν από τις επιτροπές μας. Δυστυχώ, ο εισηγητή ε, Σβέντσεν ε, δεν μπόρεσε να έρθει ε, και η κυρία Σάιφη ε, και αυτή ε, δεν μπόρεσε να έρθει, γι' αυτό λοιπόν θα τα διαβάσω εγώ τα δικά της ε, τα σχόλια η οποία γράφει και διαβάζω. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή ΝΤΕΒΕ υπογραμμίζει τα σημαντικότερα θέματα ε, και γι' αυτό ε, θα τα παρουσιάσω όλα από κοινού, αλλά παραμένω στη διάθεσή σα αν έχετε να υποβάλλετε συγκεκριμένε ερωτήσεις. Όσον αφορά στη διαδικασία, θα διαπιστώσατε ότι και η δική μα Επιτροπή και η Επιτροπή Ανάπτυξη κατάρτισαν έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 50. Ο κύριο Βένσεν αναφέρει δύο δύο θέματα ε, τα οποία δεν μπόρεσε να εντάξει στη δική μου την έκθεση και αυτό λόγω του ότι υπήρχαν ε, περιορισμοί. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και ο καθοριστικός ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είμαι λοιπόν χαρούμενη που η συνεργασία θα καταλήξει σε δύο ε, συμπληρωματικά κείμενα. Η δική μου δουλειά λοιπόν ε, υπάρχει κατ' ουσίαν στις πρώτες δύο παραγράφους ε, του σχεδίου της έκθεσης. Καταρχήν το εμπόριο και οι επενδύσεις μπορούν να αποτελούν το μέσο ε, για να υπάρξει ανάπτυξη, προκαλούν την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Βέβαια, μόνα τους τα δύο αυτά στοιχεία δεν μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την ανάπτυξη. Άρα, δηλαδή, οικονομική και τεχνική βοήθεια, όπως και παράλληλα εθνικά μέτρα, πρέπει να εφαρμόζονται η σκιώδης εισηγήτρια κατά την τελευταία συνάντησή μας ρώτησε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, προτείνει ότι είναι υπέρ του εμπορίου. Εγώ θεωρώ ότι αυτό συμβαδίζει με την πολυμέρεια. Οι διευκολύνσεις, η βοήθεια στο εμπόριο, αυτά επιτρέπουν στις αναπτυσσόμενες χώρες να επενδύσουν με τον ίδιο τρόπο όπως και οι αναπτυγμένες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλα αυτά τα εργαλεία και τα χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό και είναι εκείνη που προσφέρει τις περισσότερες ενισχύσεις. Βέβαια, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Υπάρχει η πρόταση ε, να ορίζονται, να στοχεύονται καλύτερα οι αποδέκτες θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει επίση να λαμβάνει υπόψη τη κριτήρια όπως η γενικότερη ανάπτυξη της χώρας, οι ανάγκες και οι ήδη πόροι, τη, οι πρώτε της χώρας. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στοχεύσει στην προαγωγή των τοπικών αγορών γιατί η ε, ολοκλήρωση του εμπορίου σε εμά είναι πολύ σημαντική. Η Επιτροπή ίσω σκεφτεί ε, να απλουστεύσει περαιτέρω τους ε, προτιμησιακού κανόνες προέλευσης, να δώσει τη δυνατότητα και σε μικρομεσαίους να διευκολύνει ε, την κατάσταση και να διευκολύνει το εμπόριο ε, στα ενδιάμεσα αγαθά. Και τέλος, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δουλέψει στενά με τις χώρες των αποδεκτών, γιατί έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να προτείνει πιο κατάλληλα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσφέρει περισσότερη τεχνική βοήθεια, παραδείγματο χάρη βοηθώντας τις κυβερνήσεις να βελτιώσουν τις επιχειρησιακές τους στρατηγικές ή να καθορίσουν στόχους σε άλλες σημαντικές εθνικές πολιτικές. Ένα άλλο θέμα είναι η χρηματοδότηση και η αποτελεσματικότητα των εμπορικών μέτρων. Και πάλι η απάντηση είναι περισσότερη συνεργασία, όχι μόνο ανάμεσα σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά και ανάμεσα στους διάφορους άμεσους ενδιαφερόμενους. Έτσι ώστε να μην υπάρχουν ασυνέπειες που μπορεί να είναι πολύ δαπανηρές τόσο σε επίπεδο κόστους ε, όσο και αποτελεσματικότητας να υπάρχουν κυρίως οικονομικές συνεργασίες. Εδώ βλέπουμε ότι πρέπει να κεφαλοποιήσουμε την τάση που υπάρχει και να έχουμε περιφερειακές ή τριγωνικές σχέσεις. Ε, ο σκιώδης ηγητής ε, την προηγούμενη φορά έληξε το θέμα των ΣΔΙΚ. Κατά την άποψή μου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ε, προσφέρει ενδεικτικές λύσεις, αλλά υπάρχουν και περισσότερες δυνατότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν έχει εδώ μεγάλο περιθώριο ελιγμών. Όμως, οι δύο αυτές μορφές επενδύσεων είναι απαραίτητες κυρίως αν ε, υπάρχουν συνέπειες στους προπολογισμούς από την κρίση. Εγώ ε, θα ήθελα να καταθέσω τοπολογίες και να δείξω σε ποιο βαθμό οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις ε, σε τομείς που θεωρούν προτεραιότητά τους. Ο κύριος Σόλτς αναφέρθηκε σε μορφές χρηματοδότησης στην Ευρώπη, αλλά στην Ευρώπη οι κυβερνήσεις δεν συμφωνούν για τα μέσα χρηματοδότηση. Πάντως, <clears throat> πέρα από όλα τα άλλα, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να χρησιμεύσει ε, ως ένα κίνητρο στην αγορά άνθρακα. Και τέλος θα ήθελα να καταθέσω τροπολογίες και σε κάποια άλλα ε, θέματα του εμπορίου, ε, στα εμπορικά μέτρα ή στο θέμα των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Όταν καταθέσετε τις τροπολογίες σας, μην ξεχάσετε ότι οι δύο επιτροπές έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες και γι' αυτό να εστιάσετε τις δικές σας τις προτάσεις στο εμπόριο και στις επενδύσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αυτά μας λέει η συνάδελφος κυρία Σάιφη. Και τώρα θα ήθελα να ξεκινήσει η συζήτηση. Έχουν ζητήσει το λόγο οι κύριοι Μπερέφρες, και Σόλτς. Και επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα ήθελα να σας ε, ζητήσω να περιοριστείτε στα 2-3 λεπτά. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Μιλώ εκ μέρους ε, της ε, συναδέλφου Μαρία Μπαντία που δεν μπορεί να είναι παρούσα και θα διαβάσω το κείμενο που μου έδωσε σε σχέση με αυτή την έκθεση για το εμπόριο και την ανάπτυξη βασισμένη σε επενδύσει για τι αναπτυσσόμενε χώρε μετά την εξέταση του εγγράφου που εκπώνησε η συγγήτρια και την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με εκπροσώπου του ΣΑΚΑΤΑ κατά τη τελευταία συνεδρίαση τη ΣΥΝΤΑ, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η ανακοίνωση τη Κομισιόν για το θέμα του εμπορίου και τη ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σκόπιμη γιατί επικαιροποιεί την έννοια των αναπτυσσόμενων χωρών, λαμβάνοντα υπόψη τον όλο και πιο σημαντικό ρόλο των αναδυόμενων χωρών, των χωρών BRIC. Πρέπει να ξαναθέσουμε του δεσμού μεταξύ εμπορίου, ανάπτυξη και επενδύσεων για να μπορέσουμε με επαγγελματικό τρόπο να ωφεληθούν οι δικαιούχοι και να τηρηθούν οι δεσμεύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό, όπω παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά το σεβασμό των στόχων τη χιλιετία. Σε ό,τι αφορά την έκθεση, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και να τονίσω κάποιες πτυχές που θα την κατοπτρίσω και σε κάποιες τροπολογίες. Καταρχήν, να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των εμπορικών πολιτικών και αναπτυξιακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκαιότητες ε, των χωρών δικαιούχων προσφέροντας περισσότερη τεχνική βοήθεια και πόρους σε όσους το χρειάζονται περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να επεκρινούμε να υπάρχει τεχνική βοήθεια που να μπορεί να εκμεταλλεύεται και το ανθρώπινο δυναμικό. Δεύτερον, καλύτερο συντονισμό σχεδίων και πρωτοβουλειών μεταξύ δωρητών και δικαιούχων, συνεισφέροντας σε μια καθολική στρατηγική στην, ε, στο θέμα του εμπορίου και των επενδύσεων και της ανάπτυξης και να μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πρωταγωνιστές με τη συνεργασία και την εφαρμογή. Τρίτον, να εγγυηθούμε καλύτερη συνοχή μεταξύ όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνεισφέρει στο να πετύχουμε με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο τους κοινού στόχου σε ό,τι αφορά το εμπόριο και την ανάπτυξη. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς αξιολόγησης αντικτύπου που ε, το εμπόριο συνδέεται με την ανάπτυξη. Τέταρτον, la να προωθήσουμε τις περιφερειακές επαφές για να προωθήσουμε τους δεσμούς μεταξύ εμπορίου και αναπτυσσομένων χωρών, να συμμετέχουν αναπτυσσόμενες χώρες ε, στην διαδικασία ολοκλήρωσης. Πέμπτον, να προσαρμόσουμε τους εμπορικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ευνοήσουμε την ανάπτυξη ως, όπως το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και τις ε, μονομερείς δεσμολογικές προτιμήσεις για τις ε, λιγότερο ευνοημένες χώρες, έτσι ώστε με δίκαιο τρόπο να μπορέσουν να σεβαστούν πιο αποτελεσματικά τους στόχους τους. Και θέλω να συγχαρώ τέλος την συγγήτρια για το έργο της και να της πω ότι είμαι διατεθειμένη να συνεργαστούμε για να πετύχουμε ένα ισορροπημένο κείμενο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις αυτές. Φρανσίσκο Κέλλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια. Ήδη την περασμένη φορά στην ε, προηγούμενη συζήτηση ανέφερα τα πιο σημαντικά σημεία. Δεν θα τα επαναλάβω όλα, αλλά θέλω να τονίσω ότι εδώ μιλάμε για το πώς μπορούν να βοηθήσουν ε, την ανάπτυξη των πορείων και επενδύσεις. Ε, μιλάμε για την πολιτική ανάπτυξη, μιλάμε για την ανάπτυξη των άλλων χωρών. Και αν το κάνουμε αυτό, τότε στον όλο το της αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να έχουμε κατά νου το συμφέρον της χώρας εταίρου και όχι μόνο το ευρωπαϊκό συμφέρον. Και εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς. Επίσης, όταν μιλάμε για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ε, που θα βοηθά στην ανάπτυξη, γιατί πρέπει να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη άλλων χωρών, όχι τη δική μας. Πρέπει να είμαστε σαφείς λοιπόν για το ποιο το συμφέρον μιλάμε. Η συνοχή ε, τη πολιτική αναφέρθηκε, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν είναι μόνο αρχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε γενική συνοχή των πολιτικών. Είναι σαφή και η συνθήκη τη Λισαβόνα ότι χρειαζόμαστε ε, κάτι τέτοιο για την ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι όποτε κάνουμε κάτι στο εξωτερικό και έχουμε πολιτικέ που θα εφαρμοστούν στο εξωτερικό θα πρέπει να συνάδουν με τα αναπτυξιακά συμφέροντα, θα πρέπει να συνάδουν με την καταπολέμηση της ανέχειας, ε, να οδεύουν προς την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Αυτό είναι η συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη. Είναι υποχρέωση από τη συνθήκη, από τις συνθήκες. Και το εμπόριο βεβαίως και μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη, αλλά πρέπει να δούμε και για τι είδους εμπόριο μιλάμε, προς τα ποια οδό κατευθύνεται και επίσης μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο το εμπόριο, αλλά ένα μικρό ρόλο, όχι μεγάλο ρόλο. Αλλά και πάλι πρέπει να συζητήσουμε για το ποια μορφή πρέπει να πάρει το εμπόριο αυτό και ποια μορφή πρέπει να πάρουν επενδύσει. Θέλω επομένω να ρωτήσω, να θέσω μια γενική ερώτηση, ίσως να με βοηθήσει και η Κομισιόν εδώ. Δηλαδή, για ποιο είδου επενδύσει μιλάμε, για συγχωνεύσει και εξαγορέ ε, ή για ε, κερδοσκοπικές επενδύσεις ή για παραγωγικέ και νέε επενδύσεις. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντοτε να κάνουμε μια διάκριση για το ποιο είδους μιλάμε και θα ήταν καλό να έχουμε κάποιε αποδείξει από την, κάποια στοιχεία από την Κομισιόν για τι είδου επενδύσει μιλάμε στι αναπτυσσόμενε χώρε. Δηλαδή, σε τι ποσοστό, ε, τι καλύπτουν αυτές οι επενδύσεις για τις πρώτες ύλες. Να σας πω ότι εμείς πιστεύουμε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν ε, τους ε, ε, τις εξαγωγικούς περιορισμούς προκειμένου να μπορούν να υποφελούνται και οι ίδιες από τις δικές τους πρώτες ύλες για να αναπτύξουν τις δικές τους βιομηχανίες και, αυτό, και είναι σημαντικό επίσης να υπάρχει διαφοροποίηση της οικονομίας τους. Και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω την Κομισιόν πότε σκοπεύετε να ξεφορτωθείτε αυτή την κλίμακα στους δασμούς ε, που ε, ουσιαστικά μας οδηγεί στην εισαγωγή πρώτων υλών από τις τρεις χώρες με αποτέλεσμα να μην μπορούν αυτές οι χώρες να διαφοροποιήσουν την οικονομία τους. Και αυτό που θα έπρεπε μάλλον να κάνουμε ε, θα έπρεπε να βοηθήσουμε αυτές τις ε, τρίτες χώρες ε, να σεβαστούν τους φυσικούς πόρους και να εκμεταλλευτούν αυτούς τους πόρους με υφόρο τρόπο. Και κάτι τελευταίο για τη Γεωργία. Η συγγήτρια έχει μια παράγραφο σχετικά για το θέμα αυτό είναι επίσης σημαντικό για το ποια γεωργία μιλάμε. Γιατί αν μιλάμε για τη σημερινή μορφή γεωργίας, ε, τότε το εμπόριο μας οδήγησε στο ε, να εξάγονται, παραδείγματο χάρη, πάρα πολύ φτηνά ή πολύ μετακοτόπουλου ε, σε φτωχές χώρες και υπάρχουν κάποιε δομέ που οικοδομήθηκαν εκεί και με αναπτυξή βοήθεια. Δηλαδή, ξοδεύουμε δύο φορές χρήματα. Δηλαδή, και ε, ουσιαστικά όταν εξάγουμε εμείς τα δικά μας κοτόπουλα, ε, αλλά και όταν εκεί ε, δημιουργούμε κάποιους οργανισμούς τοπικούς, δύο φορές ξοδεύουμε τέτοια χρήματα. Και θα ήθελα να αναφέρω και τα δικαιώματα διανοητικής διοκτησίας, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πιστεύουμε ότι δεν θα έπρεπε να ζητήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να σεβαστούν αμέσω τα διεθνή πρότυπα για το IPR. Το σημαντικό είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν προσβάσει τη τεχνολογία και να έχουν πρόσβαση στην ιατρική αλλά και σε άλλες ε, τεχνολογίες ε, και σε πράσινες τεχνολογίες. Δηλαδή ε, το να ακολουθούμε την αυστηρή οδό του σεβασμού των δικαιωμάτων της δεν είναι ο κατάλληλος δρόμος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλερ. Ο κύριος Σόλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κοιτάξτε και εμείς επισημάναμε την κατάσταση που ισχύει σχετικά με τις δύο αυτές εκθέσεις και επιτρέψτε μου να πω το εξής. Όταν έχουμε δύο εκθέσεις ε, οι οποίες ε, τοποθετούνται για την ίδια ε, απόφαση της Κομισιόν και ανταλλάσσουν πληροφορίες, τότε τίθεται το ερώτημα πόσο κοστίζει αυτό σε μετάφραση, σε χρόνο, δηλαδή μήπως τελικά μόνοι μας ε, δεν προβάλλουμε μια αρνητική εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τα λέω όλα αυτά γιατί ξέρετε και τις δύο εκθέσεις ε, τις ε, βρίσκω καλές και θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Σάιφη για το σχέδιο που κατέθεσε. Αυτό που ενδιαφέρει τώρα είναι κατά την άποψή μου να κατανοήσει κανείς την προοπτική της, ε, του άλλου και πώς είναι δυνατόν να υπάρξει κάποια σωστή εξέλιξη. Και τα λέω όλα αυτά έχοντας κατά νου ότι δεν ασχολούμεθα πρώτη φορά με την ε, ιστορία ε, η οποία καθορίζεται από αμοιβαία ε, δυσπιστία. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό αφορά και τις ε, γραμματείες. Το λέω αυτό λοιπόν ξεκάθαρα, διότι πιστεύω ότι με την έκθεση ή με τις εκθέσεις αυτές έχουμε την ευκαιρία να προβούμε σε διόρθωση της πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατόπιν τούτου, θα ήθελα να προσπαθήσω να διατυπώσω κάποιες ε, τροπολογίες ε, στην έκθεση. Πάντως, αυτό το είπα ήδη την τελευταία φορά, δεν θα είναι πολλές οι προτάσεις, διότι η έκθεση, κατά την άποψή μου, περιλαμβάνει πολλά και σημαντικά στοιχεία. Και σήμερα άκουσα, κύριε Πρόεδρε, ε, αυτά που μας διαβάσατε, την άποψη της κυρίας Σάιφη, όπου καθιστά σαφές που επιθυμεί να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη. Νομίζω λοιπόν ότι επισήμανε λιγάκι το θέμα της εταιρική κοινωνικής ευθύνης. Αν δούμε όμως τις τελευταίες εξελίξεις στο Μπαγκλαντές, οπωσδήποτε η ασφάλεια στη θέση εργασίας είναι κάτι το σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρουμε. Όσον αφορά τώρα τις επενδύσεις, ε, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι αναφέρεται στο εδάφιο υπαριθμών Γ. Εκεί αναφέρεται ότι οι επενδύσεις ε, δεν μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλληψη διαρθρωτικών αδυναμιών. Αλλά η ίδια η στο 4 καταλήγει σε διαφορετικό συμπέρασμα. Γι' αυτό λοιπόν ίσως ε, θα πρέπει να δούμε λιγάκι καλύτερα την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων. Τώρα, πιο κάτω που γίνεται λόγος για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Αυτό θα ήθελα να αναφέρεται περισσότερο στο κεφάλαιο βιομηχανία και όχι στις υπηρεσίες που αναφέρεται. Όσον αφορά τα EPR, θέλω να σας πω ότι κατά την άποψή μου ε, κομισιόν είναι εκείνη που φέρει την κύρια ευθύνη για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Και δεν καταλαβαίνω γιατί η ε, Κομισιόν επιμένει ε, στην κατάργηση των φορολογικών δασμών ο φόρος δεν είναι απαραίτητα προστατευτικό μέτρο, όπως αναφέρεται, αλλά ένα κλασικό ε, μέτρο άσκησης βιομηχανικής πολιτικής. Έτσι λοιπόν εμείς θα προσπαθήσουμε την έκθεση αυτή να την εμπλουτίσουμε και να συμβάλλουμε στο να ε, είναι συγκεκριμένη η έκθεση. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τη συνάδελφο κυρία Σάουιφη για αυτή την πολύ καλή έκθεση. Vielen herzlichen Dank. Herr bitte. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Είναι εξαιρετική η μοίρα του τύχη του Διεθνού εμπορίου και των επενδύσεων ε, είναι αναφεσβήτητα ένας παράγοντας ε, ανάπτυξη, αλλά θα ήθελα να αφιστήσω την ε, προσοχή σας στο ότι Ουσιαστικά αυτή η παραδοχή είναι κάπως μονομερής, ε, γιατί οι συνέπειες ε, του εμπορίου και των επενδύσεων στην πραγματικότητα είναι ποικίλε, ε, είναι αντιφατικές. Γενικά ήταν θετικός ο πολλαπλασιασμός, η αύξηση του εμπορίου τα 30 τελευταία χρόνια, γιατί γενικά είδαμε ότι αναπτύχθηκε η παγκόσμια οικονομία και αναπτύχθησαν πολλέ χώρε, αυτέ που καλούμε οι μεγάλε αναδυόμενε χώρε και είναι πολύ περισσότερε από τι BRIC. Είναι δεκάδε. Όμω ε, υπήρξαν και αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή ε, το να πολλές χώρες, αυτές που καλούμε οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Και η έκθεση το υπογραμμίζει αυτό και μας λέει ότι εφ' εξής οι προτιμησιακές συμφωνίες θα πρέπει να στοχεύουν καλύτερα δεν αρκεί να έχουμε πρωτευουσιακέ ε, συμφωνίε με την Κίνα, τη Βραζιλία ή κάποιε άλλε τέτοιε χώρε, ενώ θα έπρεπε να επικεντρώσουμε αυτή τη βοήθεια στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες που βρίσκονται σε τέλμα και μάλιστα πολλές φορές και σε ύφεση. Δεύτερον, σωστά υπογραμμίζει η συγγήτρια ότι ο κατάλληλος χώρος για την ανάπτυξη είναι επίσης να δούμε ε, σε διάφορα επίπεδα, σε υπηρετικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Και θα πρέπει να επιμείνουμε στο να ε, οργανωθεί βοήθεια με ένα τέτοιο τρόπο για να έχουμε ολοκλήρωση στα επίπεδα αυτά. Επίσης γίνεται αναφορά στα κύρια εμπόδια των συναλλαγών και αναφέρεται ότι δεν είναι δεσμολογικά τα εμπόδια αυτά και μεταξύ αυτών που μπορούμε να αναφέρουμε, κυρίως στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, είναι η ανεπάρκεια των υποδομών και ε, της οργάνωσης και της επιμελητίας και η δυσκολία να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες ασφαλείας που καθορίζουν την πρόσβαση στην αγορά των ε, πιο αναπτυγμένων χωρών των διεθνών αγορών. Η μικρή πρόσβαση και το κόστος της πρόσβασης της απαραίτητες ε, πληροφορίες. Η ανεπάρκεια του συστήματος του πιστοτικού Όλοι αυτοί είναι παράγοντες υποανάπτυξης που θα ε, έπρεπε να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη και που εν μέρη λαμβάνει υπόψη η έκθεση. Και καθώς εν μέρη λαμβάνει υπόψη η έκθεση τα θέματα αυτά, εγώ θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες να τα λαμβάνει υπόψη πλήρως. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον κύριο Ντένις Μπερέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και την συγχύτρια για την εκθεσή της. Βλέπουμε ότι υπάρχει γενικά υποστήριξη της πολιτικής που έχουμε θετήσει από την έκθεση. Έχω κάποια σχόλια και θα προσπαθήσω να απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν, ε, για την έννοια της διαφοροποίησης. Ε, υπάρχει στην έκθεση, αλλά νομίζουμε ότι θα πρέπει να δίνεται περισσότερη έμφαση. Η έμφαση στις λιγότερο αναπτυγμένες ε, χώρες, που είναι ο πυρήνας της νέας μας πολιτικής μας, είναι κάπως αδύναμη. Επίσης, ίσως και οι ευθύνε των αναδυόμενων οικονομιών θα μπορούσαν να αποσαφήνιστούν στην έκθεση. Στην παράγραφο Δέλτα, ουσιαστικά συμβαίνει το αντίστροφο, δηλαδή μπορούν ε, η ευρωπαϊκή πολιτική να, μπορεί, η ευρωπαϊκή πολιτική να συμπληρώσει τι εθνικέ πολιτικέ και όχι το αντίστροφο. Και αυτό έχει να κάνει με τη τεχνική βοήθεια. Εμεί είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε τεχνική βοήθεια, αλλά φυσικά εξαρτάται και από τι χώρε εταίρους να αποφασίσουν αν τη χρειάζονται και να τη ζητήσουν. Δεν μπορούμε να του την επιβάλλουμε. Παράγραφος 5 Υπάρχει ένα μικρό, μακρύς κατάλογος στόχων και είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι περισσότεροι από αυτού του στόχου πρέπει να επιδιωχθούν μέσω εθνικών πολιτικών από τι αναπτυσσόμενες χώρε αυτέ καθ' αυτέ. Παραγραφός 6 αναφέρεται στο θέμα του κατακεφαλήν εισοδήματο ω κριτήριο για τη βοήθεια. Οι περισσότερες προτεραιότητες μας ε, κατευθύνονται τώρα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και έχουμε τρία κριτήρια το κατακεφαλή και ε, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την, το να βάλει το χαρακτήρα σε εξωτερικούς, εξωτερικούς κραδεσμούς. Όμως ε, το κριτήριο του εισοδήματος κατά έχει γίνει αποδεκτό ως ένα σχετικό κριτήριο. Παράγραφος 15 για τους κανόνες καταγωγής. Να υπενθυμίσω ότι μεταρρυθμίσαμε τους ε, κανόνες γενικευμένου συστήματος προτιμήσεων για την καταγωγή, τους απλοποιήσαμε, τους χαλαρώσαμε και τώρα του χρησιμοποιούμε ως δείγμα για τις ε, διάφορες συμφωνίες, συμφωνίες ελευθερίου εμπορίου, ε, τις EPAs κτλ. Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 16, να αποσαφηνίσω ότι ναι, θα παρουσιάσει συχνά σε εκθέσει κομισιών ε, για τα αποτελέσματα του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων σύμφωνα και με τις απαιτήσει του άρθρου 40 για τις IPAs. Νομίζω ότι η Κομισιόν ε, έλαβε υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε τρεις τέτοιες συμφωνίες που εφαρμόζονται τώρα και μία στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένης μίας της Αφρικής. Η Κομισιόν ε, θεωρεί ότι η διάβρωση είναι αναπόφευκτη, αλλά θα λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα των χωρών και, και των ευαίσθητων προϊόντων στις διαπραγματεύσεις για τις FTA. Ε, τώρα για την ευελιξία νομίζουμε ότι έχουμε δείξει αρκετή, αλλά για να ε, πάμε στο τελικό στα διαπραγματεύσεων δεν χρειάζεται τώρα ευελιξία, αλλά πολιτική βούληση. Και για την παράγραφο 18 να σας πω ότι σε αυτή την έκκληση που ευθύνεται της Κομισιόν. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό αντιμετώπισε και κάλυψε και η ανακοίνωση της Κομισιόν για τις επενδύσεις. Νομίζω ότι εξαρτάται και πόσε επενδύσει προσελκύει μια χώρα, αλλά αυτό εξαρτάται από το νομικό περιβάλλον, τι τοπικέ συνθήκε. Νομίζω ότι διότι εμπορική πολιτική, σκοπεύουμε περισσότερο, σκοπεύουμε περισσότερο σε επενδύσει στι ε, υποδομές ε, σε ό,τι αφορά τώρα την κλιμάκωση της, ε, των δασμών. Αυτό δεν αφορά τις χώρες που είναι σε μεγαλύτερη ανάγκη. Εκεί δεν υπάρχουν μάλιστα και καθόλου δασμοί. Στις λιγότερα αναπτυγμένες χώρες έχουμε πολύ χαμηλούς δασμούς. Ανάλογα με το αν οι χώρε είναι δικαιούχοι του γενικού συστήματο προτιμήσεων ή ανήκουν σε μια συμφωνία EPA FTA. Και δεν νομίζουμε ότι το θέμα των δασμών και με το διάβρωση ε, το ένδεσμο αυτό είναι το πλέον σημαντικό, αλλά όπω και να έχει το αντιμετωπίζουμε. Σα ευχαριστώ. Και δεν ξέρω αν συνάδελφο από την θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις αυτές. Υπάρχουν σχόλια ή παρατηρήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Αν όχι, τότε να σας υπενθυμίσω ότι η κατάθεση των τροπολογιών πρέπει να γίνει μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου, τις 12 και 24 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ και να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο, το 14. Έχουμε την ενδιάμεση συμφωνία που θεσπίσει πλαισίου συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ κρατανατολικής και Μεσημερινής Αφρική και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στις 3 του Οκτωβρίου είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων με τους πρεσβευτές των τεσσάρων χωρών με τις οποίες έχει συνάψει αυτές ε, τις συμφωνίες με ο Σεϊχέλης, Μαδαγασκάρη και Ζιμπάμπουε και τώρα εξαρτάται από τα μέλη της Επιτροπής μας να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν. Και θα δώσω το λόγο στον εαυτό μου γιατί είμαι εισηγητής. Συνάδελφοι, να πω καταρχάς ότι ήταν καλή ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των τεσσάρων ε, χωρών που αφορά η συμφωνία αυτή. Οι χώρες αυτές ήθελαν ε, βεβαίως να συναυθεί αυτή η συμφωνία εταιρικής σχέσης και οικονομικής συνεργασίας. Θα προσπαθήσω εδώ να απηχήσω τα πλεονεκτήματα και τα μενεκτήματα της ε, συμφωνίας αυτής από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ενδιαφερόμενων χωρών στην έκθεσή μου. Νομίζω ότι η έγκριση της ε, σχετικής συμφωνίας εταιρική σχέσης είναι ένα θετικό βήμα. Θα ήθελα να ακούσω τις παρατηρήσεις σας, ε, εάν έχετε κάτι να πείτε, κυρία Κέλλερ. Ευχαριστούμε πολύ, για την έκθεση και για την υποβολή τη. Συζητήθηκε και στην προηγούμενη Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Εγώ δεν ήμουν, αλλά άκουσα ότι ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα. Έχω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις κυρίες, για την αιτιολογική έκθεση. Στην πρώτη σελίδα λόγου χάρη λέτε οι νέες αυτές συμφωνίες θα ε, στηριχθούν από την αναπτυξική πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύσουν τις δυνατότητες παραγωγής ε, του, των χωρών αυτών. Λέτε δηλαδή ότι θα ενταθεί η αναπτυξιακή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσατε να διευθύνσετε τι αύξηση θα είναι αυτή. πώς θα βοηθηθούν οι χώρες αυτές, ποιοι είναι οι τομείς που θα ενισχυθούν. Αυτό θα ήταν σημαντικό να το γνωρίζουμε. Επίσης, για το θέμα της περιφερειακής ε, ολοκλήρωσης. Συμφωνώ με το στόχο να υπάρξει περιφερειακή ολοκλήρωση, αλλά δεν είμαι βέβαιη πως αυτή η, ενδιάμεση έκθεση μπορεί να βοηθήσει, η ενδιάμεση συμφωνία μπορεί να βοηθήσει. Όπως είπατε και ο ο ίδιος, μόνο Μερικά από τα 11 κράτη έχουν ε, αποφασίσει να συνάψουν συμφωνία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και διαφορετικέ απόψει εκεί. Σημαντικό είναι να δούμε αν τα 11 κράτη θεωρούν ότι υπάρχει βελτίωση για την περιφερειακή ολοκλήρωση μέσω των συμφωνιών αυτών. Διότι εμεί μπορεί να επιδιώκουμε την περιφερειακή ολοκλήρωση, αλλά τα κράτη θα πρέπει να δούνε πώ θα εκτελεχθεί αυτή η περιφερειακή ολοκλήρωση. Και για την ώρα, αυτά που έχω ακούσει από του εκπροσώπου των ε, ενδιαφερομένων κρατών έχουν ε, ανησυχίες και αμφιβολίες για το πώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν την περιφερειακή ολοκλήρωση. Ιδίω την κοινή αγορά στην ε, Νότια Αφρική. Ίσως θα θέλατε να το σχολιάσετε. Επίσης, έχω και μια ερώτηση για την επαρκή προστασία της ε, βιομηχανίας Ε, τι εννοούμε με, την, με τον όρο επαρκή προστασία. Επίση, κάποιε χώρε έχουν αρχίσει να υλοποιούν μέρη τη συμφωνία από το Μάιο. Δίκιο νομίζω έχετε. Εάν, ε, αλλά θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να συναγάγουμε συμπεράσματα ήδη από τώρα. Γιατί καλό θα είναι να δούμε πώς οι συμφωνίες αυτές υλοποιούνται στην πράξη και τι είδου διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από τη συμφωνία και να δούμε και τι επιπτώσεις υπάρχουν. Και ίσως ένα τελευταίο ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, εγγύησεις. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι νόμοι, τα νομοθετήματα ή τέλος πάντων οι κανονισμοί για τις τέσσερις χώρες που μπορούν να αναχαιτήσουν την απότομη των εισαγωγών και εάν υπάρχουν οι ανάλογες θεσμικές ε, εγγύησεις Τέλος, οι χώρες αυτές έχουν τι τεχνικές δυνατότητες να εφαρμόσουν τα μέρη της συμφωνίας και είναι και πολιτικό το ζήτημα, αλλά μιλάμε για οικονομικούς δεσμούς πια με τις χώρες αυτές και ευρωπαϊκές εταιρείε θα πάνε στις χώρες αυτές. Πώ ακριβώς θα διοργανωθεί όλο αυτό. Αυτές είναι ερωτήσει μου και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ θα γίνει. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μουσκαρντίνη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω Ντανιέλ για αυτήν την ε, τόσο λεπτομερή και συνοπτική πλήρη έκθεση. Να θυμίσω την ανάγκη να δίνουμε διαρκώς όλο και μεγαλύτερη προσοχή ε, στη σχέση μας με την Αφρική. Η Αφρικανική Ήπειρος εκπροσωπεί έναν από τους ε, πιο σημαντικούς εταίρους μας. Αν και τίνουμε να το αμελούμε με, τον, με τα χρόνια, ιδίω πρόσφατα, η έντονη κινέζικη παρουσία στην Αφρική, η οποία αγόρασε εκατομμύρια εκατομμυρίων εκτάρια, αυτή τη στιγμή συνοδεύεται και από έντονη βραζιλιανική παρουσία. Από εμπορικής λοιπόν και παραγωγικής σκοπιάς Βλέπουμε πολιτική των χωρών αυτών στην ε, Αφρικανική Ήπειρο να μην πω ότι είναι υπεραλιστική επιθετική, αλλά σίγουρα προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Θέλουμε λοιπόν συμφωνίε χρήσιμε και για του Αφρικανού και για την ευρωπαϊκή πλευρά και ε, προ αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να προχωρήσουμε για να γίνουν πιο εντατικέ οι σχέσει και πιο σταθερά τα προγράμματα που θα μπορούσαν να προσδώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνατότητες να γίνει ένας σοβαρός συνομιλητή. σοβαρός συνομιλητή της Ευχαριστώ. Thank you very much, Paul Murphy, please. Ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, έκθεση. Ε, κοιτάξτε, μετά από τις ε, τελευταίες συζητήσεις που είχαμε με τους πρέσβεις των χωρών, αισθάνομαι ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτή τη ε, γλώσσα της ε, περιφερειακής ολοκλήρωσης. Ε, Κοιτάξτε, αυτή η συμφωνία, η διάμεση που υπογράφηκε, καταδεικνύει ότι ε, δεν διευκολύνεται η περιφερειακή ολοκλήρωση. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση η περιφερειακή ολοκλήρωση ε, καθίσταται ε, πολύ πιο δύσκολη ανάμεσα στις άμεσα ενδιαφερόμενες χώρες. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά στη μέθοδο με την οποία διεξάγονται αυτές οι διαπραγματεύσεις όπου ε, όλες οι ενώσεις, ε, οι εκπρόσωποι της Αφρικανικής Ένωσης ε, των ΜΚΟ δείχνουν ότι η Κομισιόν διεξάγει τις διαπραγματεύσεις με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο, δηλαδή αγνοεί τις ανάγκες και τις ανησυχίες των χωρών και σπάει τη Συμφωνία Κοτονού και ακολουθεί δική της, ε, το δικό της το θεματολόγιο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και το τρίτο αφορά στη φύση της ε, συμφωνίας. Ε, οι χώρες ίσα απαιτούν την αναθεώρηση να μπορούν να μειωθούν οι δασμοί. Εδώ υπάρχει ένα μικρό χρονικό διάστημα, τα 15 χρόνια, ενώ η, στην η απελευθερωποίηση λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν και εξαιρέσεις ενό 20% και σε ορισμένε χώρες όπως είναι η Ασία, ακόμα και το 98% της ε, απελευθέρωσης. Αυτό θα είχε ε, πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις εσωτερικές ε, αγορές. Προφανώς η όλη διαδικασία είναι αρκετά διευρυμένη αλλά η Οικονομική Επιτροπή για την Αφρική έχει καταθέσει αρκετές ε, μελέτες όπου όλα αυτά θα είχαν ε, την υπονόμευση της ε, κοινωνικής συνοχής. Δεν νομίζω ότι η Κομισιόν έχει απαντήσει σε όλες αυτές τις ανησυχίες και γι' αυτό διαφωνώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή πολλά τέθησαν προς την Κομισιόν θα ήθελα να δώσω και το λόγο για να απαντήσει σε όλες αυτές τις ε, ερωτήσεις. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τον εισηγητή και τα διάφορα μέλη που έθεσαν ερωτήσεις. Θα ήθελα να πω το εξής όσον αφορά στο θέμα που έχει σχέση με τις ε, διατάξεις ε, προστασίας και διαφύλαξης, ε, δηλαδή να ανασταλεί η προτιμησιακή συμφωνία στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, κίνδυνος βλάβης μάλλον, πρόκληση ζημιάς. Ε, εδώ λοιπόν υπάρχει αυτό που αποκαλούμε και τα διμερεί μέτρα προστασίας εμείς θεωρούμε ότι εδώ έχουμε ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο. Άρα δηλαδή δεν σημαίνει ότι το χρησιμοποιούμε το μέτρο αυτό, αλλά το πλαίσιο είναι σαφές ε, και όπως βλέπετε το άρθρο είναι αρκετά μακροσκελές. Όχι για να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά για να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να εφαρμοστεί και ότι οι συνθήκε είναι ξεκάθαρε, οι όροι είναι ξεκάθαροι. Οι ε, τέροι μας έχουν την δυνατότητα να επικαλεστούν ένα τέτοιο μέτρο σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο και εμεί ε, θεωρούμε ότι όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή μπορούμε να την ε, προσφέρουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήθελα να αναφέρω. Υπάρχει λοιπόν και ένα συγκεκριμένο ερώτημα που αφορά στην στήριξη της συνεργασίας και επ' αυτού θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στο συνάδελφο μου από την Europaid. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν θα έχω ολοκληρώσει βέβαια εγώ. Θέλω επίσης να πω ότι επιπρόσθετα στην ρήτρα προστασίας ε, υπάρχει και μία ρήτρα που αφορά για την εργασία, για την νεόκοπη βιομηχανία, τις ε, νέες επιχειρήσεις. Επίσης, όσον αφορά και τη συνεργασία που μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τη λειτουργία της ε, συμφωνίας και εδώ πάω στο θέμα των επιπτώσεων από αυτή τη ε, συμφωνία. Βεβαίω είναι πάρα πολύ νωρί για να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε κάποιες επιπτώσεις. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι ο Μαυρίκιος άρχισε τον περιορισμό δασμών που είχε δεσμευτεί και άλλες χώρες έχουν δεσμευτεί, αλλά ακόμα δεν έχουν προβεί σε αυτές τις ε, περικοπές. Και κάτι άλλο οι θεσμοί που αναφέρονται στη συμφωνία έχουν αρχίσει να λειτουργούν. Άρα δηλαδή πλέον η συνεργασία έχει ύπαρξη. Είχαμε μία συνάντηση της Επιτροπής ΥΠΕ, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής για τη Συνεργασία στα Δασμολογικά. Και αν μου επιτρέπετε να μπω και σε λεπτομέρειες, υπάρχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα από αυτές τις ε, συναντήσεις. Οι εταίροι ίσα ε, έχουν πάρει αυτό που αποκαλείται αυτόματος εξαιρέσεις ε, για την προέλευση ενός βασικού προϊόντος όπως είναι ο τόνος. Αυτό από την 1η Ιανουαρίου. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα που επιτύχαμε. Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην Αφρική. Υπάρχει ένας συγκεκριμένο τρόπος, ενδιάμεσος, που μπορούμε να το επιτύχουμε. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Γιατί ετέθη από πολλούς και βρίσκεται το θέμα αυτό στην καρδιά όλου αυτού του εγχειρήματος. Αυτό που έχουμε είναι μια ενδιάμεση προσωρινή συμφωνία με μια σειρά κρατών. Και όπως είπε και ο διευθυντής μου, όταν, είπε, όταν ήρθε στην πρώτη συζήτηση, να λέμε ότι αυτό θα ήταν ε, το τέλειο, αυτό ε, είναι λάθος. Αλλά και να λέμε ότι παρεμποδίζει την περιφερειακή ολοκλήρωση Αλλά και αυτό δεν είναι αλήθεια. Εκείνο το οποίο έχουμε εδώ είναι ένα πλαίσιο για συνεργασία ανάμεσα σε αυτές τις χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πλαίσιο έτσι ώστε και αυτές να συνεργάζονται στενότερα μεταξύ τους. Βλέπουμε λοιπόν πως ε, η δική μας ε, η δουλειά, αυτή που έχουμε ξεκινήσει εμείς, δηλαδή το να υπάρχουν τα σωστά εργαλεία για τα δασμολόγια, για τους δασμούς γενικότερα. Αυτό μπορεί να είναι τεχνική δουλειά, αλλά στηρίζει την διαδικασία της ολοκλήρωσης. Αν θέλετε κύριε Πρόεδρε, μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, αλλά νομίζω αυτή μπορεί να είναι η πρώτη μου απάντηση και θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στη συνάδελφο για να μιλήσει για την ε, συνεργασία. Καλημέρα σας, λέγομαι Ιρένη Τζεριμπάλντι και εργαζόμαι στη Γενική Διεύθυνση για την Απτυξιακή Συνεργασία. Καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, αξιότιμο βουλευτή που ρώτησε για την ανάπτυξη, γιατί αυτό μας επιτρέπει εφενός να νεώσουμε τη δεσμευσή μας ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ε, υποστηρίξουμε την εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Σύμπραξης και επίσης να σας ενημερώσω και για το τι κάνουμε. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία φέτος το Μάιο. Και όπως επίσης αναφέρεται στην έκθεσή σας, ε, υπάρχει ένα κεφάλαιο ανάπτυξης της αναπτυξιακής συνεργασίας ε, που καλύπτει και τη συνεργασία με τις ε, χώρες εφαρμογής και επίσης προβλέπεται η σύσταση μιας ε, κοινή αναπτυξιακής επιτροπής η οποία θα αναφέρεται ως κοινή επιτροπή ΙΠΑ. Επίσης, ε, να σας πω ότι στις 19 Οκτωβρίου συζητήσαμε αυτή την Επιτροπή και κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής ε, κάναμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και συμφωνήσαμε για την αναπτυξιακή πλευρά της συμφωνίας. Καταρχήν, μας ρωτήσατε τι ακριβώς κάνουμε σε σχέση με την αύξηση ή τη μείωση. Εξετάσαμε τι είχαμε ε, σε ό,τι αφορά στα εφιστάμενα προγράμματα και επίσης ε, ε, συγκεντρώσαμε μία σειρά μέτρων που είναι σήμερα ακόμη ανοιχτά και μέσω του EDF και του DCI και μιλάμε για 830 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι διαθέσιμα σήμερα υπό τη μορφή πρωτοβουλειών και κατόπιν αναφέρθηκε πήκαμε συγκεκριμένα στο εξή. Καλέσαμε τη χώρα να προτείνει δράσεις αναλόγως με τις ανάγκες της. Στα προγράμματα που υπάρχουν, Και σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε περιφερειακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται ε, από το περιφερειακό πρόγραμμα για τον Ειρηνικό Κένο και την Νότια Αφρική. Έχουμε το ε, πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης που έχει ως στόχο να υποστηρίξει χώρες για τη ευκολήση του εμπορίου, την ανάπτυξη του εμπορίου, για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα υποξήριξη των κρατών μελών ε, για ε, να εφαρμόσουν την απελευθέρωση του εμπορίου και έχουμε 17 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα αυτό. Πολύ λίγα έχουν χρησιμοποιηθεί και καλέσαμε τις χώρες να προτείνουν δράσεις ε, για να έχουν ένα κονδύλι υπό το πρόγραμμα αυτό. Ακριβώς για να υποστηρίξουμε τις χώρες που αντιμετωπίζουν την πρόκληση εφαρμογής μιας τέτοιας συμφωνίας. Αυτό ως παράδειγμα, αλλά έχουμε και άλλα προγράμματα υπό τα περιφερειακά ταμεία ή ε, βάση διμερών προγραμμάτων που ήδη υφίστανται αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ένα πρόγραμμα υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα, απασχόληση και περιφερειακό εμπορίο για τη Μαδαγασκάρη, 8 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αυτή τη ε, στιγμή το συζητούμε και το διαμορφώνουμε με την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης. Έτσι λοιπόν δεν περιμένουμε Επίσης, ε, επειδή υπήρχαν συγκεκριμένες ανάγκες που πρότειναν οι χώρες, ε, προστιμούμε να ε, αναπτύξουμε κάποιες εκστρατείε ευαισθητοποίησης για τις επιχειρήσεις και ζητήσαμε από τις χώρες να προετοιμάσουν μια αξιολόγηση των αναγκών που έχουν και σχετίζονται άμεσα με τη συμφωνία, γιατί Σήμερα είμαστε στο στάδιο προγραμματισμού του N10, του EDF, του Αναπτυξιακού Ταμείου λοιπόν και θέλουμε να εντάξουμε στον προγραμματισμό μας σε αυτές τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής Θα εντάξουμε λοιπόν τις χώρες αυτές εκεί, το επόμενο έτος θα ξανασυναντηθούμε. Αυτά κάνουμε μέχρι τώρα. Απλώς ήθελα να καθησυχάσω τις Επιτροπές ΣΥΝΤΑ και ε, δυστυχώς βέβαια δεν μπορούν να μας ακούσουν, αλλά ότι θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε αυτές τις χώρες για την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας Οικονομικής Συντερικής Σχέσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Ως ε, εισηγήτρια ε, θεωρώ ότι αναφερθήκατε σε πολλά θέματα, αλλά βέβαια δεν ε, εξαλείψατε τις ανησυχίες όλες, όλων των συναδέλφων. Για να προχωρήσουμε όμως, ε, θέλω να πω το εξής. Η καταληκτική προθεσμία είναι 28 Νοεμβρίου, 12 η ώρα, και η, για την κατάσταση τροπολογιών και η ψηφοφορία θα γίνει το Δεκέμβριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το σημείο υπαρθμών 16 έχει διαγραφεί. Πάμε στο επόμενο θέμα ε, στις δραστηριότητες της εποπτικής ομάδας. Και να σας πω ότι στις 7 Νοεμβρίου είχαμε μία συντακτική συνάντηση της ομάδας ελέγχου για τις εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία. Και χτες οι συντονιστές αποφάσισαν ότι οι, οι ομάδες αυτές για τις σχέσεις με την Ταϊβάν, την Χιλή, την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία, οι ομάδες αυτές ελέγχου ε, θα πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν κατά τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Δεν ξέρω αν κάποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο. Αν όχι, θα ήθελα παρακαλώ να περάσουμε να διακόψουμε και θα επανέλθουμε στις